Ladies Παρακαλώ καθίστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Λυπάμαι πολύ για τη μικρή ε, καθυστέρηση. Οφείλεται στην ε, κυκλοφοριακή συμφόρηση στις Βρυξέλλες σήμερα. Και ελπίζω ε, εξ αυτού να έχουν καθυστερήσει και άλλα μέλη που δεν είναι παρόντα, όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε δύο Άκρο ενδιαφέροντα σημεία στην ημερήσια διάταξη τα οποία έχουμε διοργανώσει σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι μια παρουσίαση της μελέτης που ζητήθηκε και από την αντιπροσωπεία. Χαρά μου λοιπόν να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ανατολική Ασία και το ΕΖΙΑΝ, τον κύριο Μπουτεκόφερ, θερμό καλωσόρισμα στον κύριο Μπουτεκόφερ. Το θέμα της μελέτης είναι οι προκλήσεις της ελευθερίας των θαλασσών και αντιπαλότητας της θάλασσες ε, της ε, Ασίας θα παρουσιαστεί από τον αντινάβαρχο Πάτρικ Κεμπράρ. Τον καλωσορίζουμε θερμά, σας καλωσορίζουμε θερμά κύριε Ναύαρχε. Είναι ερευνητής στο Ίδρυμα Στρατηγικών Ερευνών που εδρεύει ε, εις Παρισίους αυτή η συνεδρίαση της ΣΕΝΤΕ που διεξάγεται χτες και σήμερα είναι αφιερωμένη βασικά στα θέματα ασφαλείας στην Ασία, στην ε, Νοτιοανατολική Ασία. Χτες είχαμε την ε, ακρόση, η οποία ακρόση ήταν αφιερωμένη στις πολιτικές στη νότια και νοτιοανατολική Συνική θάλασσα. Συζητούσαμε τη μεταρρύθμιση της πολιτικής ασφαλείας και αμήνης της Ιαπωνίας και σήμερα έχουμε τη μελέτη αυτή η οποία αναφέρεται σε παρόμοια θέματα αλλά ίσως με μια ευρύτερη ε, επισκόπηση χωρίς να χρονοτριβήσω να ζητήσω τον κύριο Μπουτεχόφερ αν θέλει να μιλήσει, αν δεν θέλετε. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον αντινάβαρχο, τον κύριο Πατρίκ Χελμπράντ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε που με καλωσορίσατε και που με καλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Για να κάναμε εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα θα ήθελα να αναφερθώ στις γεωστρατηγικές θεωρίες ε, που φέρνουν σε παράθεση τον Μάκεντα και Σπίκμαν. Η πρώτη θεωρία τονίζει τη σημασία της ε, ενδοχώρας της, ε, με, τονίζοντας τη Γερμανία και τη Ρωσία και η δεύτερη θεωρία την ισχύ των θαλασσών με αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη ΣΥΠΑ ε, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρετική ισχύ και τον έλεγχο της παράκτιας περιοχής και του ειρηνικού. Ε, όσον αφορά το θέμα, η Ευρασία είναι πάρα πολύ σημαντική στατικικά και αυτό ήταν ο στόχος της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Σοβιετική Ένωσης. Η Κίνα στο όραμα του Σπίξμαν είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα κομμάτι της περιφέρειας του ειρηνικού και αυτό ίσχυε στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά δεν ισχύει σήμερα. Η Κίνα μπορεί να θεωρηθεί σαν υπηρετική και θαλάσσια δύναμη με την εξαίρεση της περιορισμένης της πρόσβασης στα ύδατα των θαλασσών. Και ξανά βλέπουμε σήμερα μία διαμάχη μεταξύ της υπηρετικής ή μη υπηρετικής ε, ισχύως δύναμης και μίας θαλάσσιας δύναμης ε, που προσπαθεί να ελέγξει αμφισβητούμενη περιοχή θαλάσσια λόγους. Λοιπόν, η βασική αρχή των συγγραφέων είναι ότι ο ε, ούγκλος ήταν ότι πρέπει να προστατευτεί η ελευθερία της θάλασσας, ο πλούτος βασίζει σε οικονομικές συναλλαγές που κυρίως διέρχονται οι συναλλαγές μέσω των γραμμών θαλασσίων μεταφορών. Λαμβάνοντας λοιπόν, κρατώντας ανοιχτές αυτές τις διαδρομές της διόδου αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους φορείς, ε, θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς. Σε μερικές δεκαετίες η Κίνα έγινε η δεύτερη οικονομία στον κόσμο και μια στρατηγική δύναμη αυξάνοντας ε, το δυναμικό που έχει το θαλάσσιο ε, όσον αφορά εμπορικές μεταφορές και το ναυτικό, το πολεμικό. Εξαρτάται λοιπόν από την αύξηση της οικονομίας εξαρτάται από τις θάλασσες που είναι ημίκλειστες αυτές που τις περιβάλλουν με ε, νερά και με στενά από τα οποία πρέπει να γίνει διέλευση για να βγουν τα εμπορεύματα στον ωκεανό. Έτσι λοιπόν η Κίνα προσπαθεί να χαλαρώσει το όλο αυτό στενό πλαίσιο το οποίο έχει περικλειστεί και ε, έχει αυξανόμενα στατηγικά συμφέροντα προσπαθώντας να αποκτήσει την πρόσβαση στον Ινδικό ωκεανό και τον ε, Ειρηνικό ούτως ώστε να εξασφαλίσει τις θαλάσσιες οδούς ε, επικοινωνίας και μεταφορών. Ο βορειοδυτικός ειρηνικός ε, αποτελεί ε, την λογική επέκταση της ζωτικής ζώνης της, της Ινικής θάλασσας. Έχοντας μια, θαλά, μια ναυτική παρουσία στην περιοχή, μπορεί η Κίνα να ασκήσει πιέσει στους αντιπάλους της, ενδεχόμενους αντιπάλους, και να διοργανώσει εις βάθος την άμυνά της. Την τελευταία δεκαετία η, ο λαϊκός στρατός της Κίνας, το ναυτικό της Κίνας έχει εντατου, τι α, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητε πέρα από τις πρώτες αλυσίδες ε, νήσων από πλευράς Πεκίνου η, η θάλασσα της Νοτολικής ε, Κίνας μέσα στις, ε, τη γραμμή με, τη διακεκομένη είναι αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της οπότε εξασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοεία των δικών της ε, σκαφών θεωρείται δεδομένο. Κάτι όμως που δεν ισχύει για όλες τις χώρες. Η Κίνα έχει ε, δημιουργήσει διάφορες πολιτικές που παρακολουθούν ή περιορίζουν δραστηριότητε ξένων σκαφών που σε αυτή την περίπτωση είναι μη κινέζικα αλευτικά σκάφη. Στον Ινδικό ωκεανό το Πεκίνο έχει επενδύσει σε μια λυσίδα λιμένων στον Ινδικό ωκεανό που αποκαλείται η αλυσίδα των μαργαριταριών. Από το Δεκέμβριο του 2009 το κινέζικο ναυτικό έχει μια συνεχή ναυτική παρουσία στο κέρας της Αφρικής με δύο πολεμικά πλοία και ένα πλοίο εφοδιασμού για να αντιμετωπίσει την πειρατεία και να προστατεύσει τα εμπορικά πλοία της Κίνας προσπαθεί να βρει εγκαταστάσεις λιμενικές στην περιοχή και γι' αυτό υπέγραψε συμφωνία με το Τζιμπουτί όπου εκεί η Κίνα οικοδομεί ε, την πρώτη της στατιωτική εγκατάσταση για την Ινδία. Αυτή η στατηγική της αλυσίδας των ε, μαργαριταριών έχει γίνει μια πηγή ανησυχίας δημιουργώντας το συνέστημα ότι περικυκλώνονται οι χώρες από την Κίνα λόγω της θέσεως που έχουν τα λιμάνια και τις ειδικέ σχέσεις που έχει η Κίνα με το Πακιστάν. Τα κινέζικα συμφέροντα έφτασαν στη Μεσόγειο πρώτα απ' όλα για εμπορικού σκοπούς και πρόσφατα με ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού. Έχει δημιουργήσει πλατφόρμα στο, για εμπορευματοκιβώτια στο Port Said στην Αίγυπτο και το λιμάνι του Πειραιά είναι σε κινέζικα χέρια. Στην Αργερία μια κινέζικη εταιρεία κατασκευάζει ένα νέο λιμάνι και ε, τελικά ε, το αλγερινό ναυτικό αγόρασε κινέζικα σκάφη. Παρόλο που οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση, επίσημα έχει δημιουργήσει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων γύρω από τι ακτέ των Ηνωμένων Πολιτειών και έδωσε και στις άλλες χώρες την ελευθερία της ναυσιπλοείας εντός αυτής της ζώνης. Έκτοτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχώς επαναλάμβανε το, το κεντρικό χαρακτήρα της ελευθερίας της ναυσιπλοείας για την θαλάσσια πολιτική της χώρας και θα εξακολουθεί να επιδιώκει την πρόθεση εθνικών συμφερόντων στην νότια συνική θάλασσα βάσει αυτής της τοποθέτησης. Οι Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποκλίνουσες απόψεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η ασυμβατότητα των θέσεών τους είναι μια πηγή εντάσσεων στην ε, νότια συνική θάλασσα. Όπως η Ιαπωνία και άλλες χώρες της περιοχής, η Κίνα έχει εκφράσει ανησυχία για την ιδέα ότι ξένα πολεμικά σκάφη θα μπορούν να ε, δραστηριοποιούνται και να επιχειρούν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ε, ζώνης. Η στάση του Πεκίνου όσον αφορά την ελευθερία της αυσιπλοείας στη νότια συνική θάλασσα παραμένει αμφίσιμη και πολλά εξαρτώνται από την ε, ερμηνεία του καθεστώτος των αξιώσεών της των θαλασσίων στη διακεκομένη γραμμή που έχει, στα σύνορα, στα όρια που έχει θεσπίσει. Ε, η Ουάσιγκτον έχει ευρύ ορισμό ότι Άγκλος θεωρώντας ότι οι στρατιωτικέ δραστηριότητε επιτρέπονται σε οποιαδήποτε αποκλειστική οικονομική ζώνη όπως την ανοιχτή θάλασσα. Σήμερα με την επέκταση των δραστηριοτήτων στην υφαλοκρηπίδα σε πολλές αποκλειστικές οικονομικές ζώνες αυτή η ερμηνεία θα μπορούσε να συζητηθεί. Και οι δύο απόψεις αυτών των χωρών είναι νομικώς εύθραυστες η άποψη της Κίνας λόγω της πρόσφατης απόφασης του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών διότι δεν έχει ακόμα η χώρα αυτή κυρώσει την σύμβαση. Το 2011 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επανεξισορροπήσουν στην θέση του σε παγκόσμιο επίπεδο και στη θέση τη Ασία και του Ειρηνικού. Βασική προτεραιότητα στρατηγική ήταν η ενίσχυση τη συμμαχία με την Ιαπωνία και με την Νότια Κορέα, αναπτύσσοντα μια ισχυρή εταιρική σχέση με την Ινδία και την Ινδονησία, ενισχύοντα τις, περιφερειακού τους περιφερειακούς όπως είναι ο Έζιαν, όλο ιδιαίτερο και δημιουργώντας επικοδομητική σχέση με την Κίνα σύμφωνα με τη θέση που έχει μεταξύ άλλων χωρών διπλωματικά, στατιωτικά και οικονομικά. Η προτεραιότητα του Προέδρου Ομπάμα ήταν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον τέτοιο, ούτως ώστε μια στατιωτική αντιπαράθεση ε, γίνεται κάτι ασύλληπτο, απίθανο. Όμως εντός της αμυντικής κοινότητας των ΗΠΑ ε, υπάρχουν δύο αντίθετες τάσεις. Η πρώτη θεωρεί ότι μια σύγκρουση με την Κίνα είναι κάτι δυνατόν, αν, όχι αναπόφευκτη και θα πρέπει να προετοιμαστεί καταλήλως η χώρα, είπα. Η άλλη θεωρία είναι ότι μια αυξανόμενη, αναπτυσσόμενη οικονομία σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη αυτομάτως συμπεριλαμβανομένη της στατιωτική ισχύω. Και από πλευράς των ΗΠΑ η προσπάθεια συγκράτησης αυτής της επέκτασης είναι κάτι ε, κανονικό και σύνηθες, αλλά θα πρέπει αντιπαράθεση να παραμείνει στα πεδία τα πολιτικά και οικονομικά. Η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί το Πεκίνο σαν μια βασική πρόκληση ε, έναντι των συμφερόντων της χώρας στην Ανατολική Ασία και ακολούθησε μεικτή στρατηγική επανεξισορρόπησης και συγκράτησης της ανάπτυξης και της επιρροής της Κίνας ε, και της στατικής θέσης στην περιοχή. Από πλευράς Κίνας, η Ουάσιγκτον έχει οθετήσει εχθρική στρατηγική συγκράτησης και ε, οι ένοπλε δυνάμει των ΗΠΑ είναι σημαντική απειλή όσον αφορά την εθνική ασφάλεια τη ε, Κίνα και στρέφεται 100 συμφερόντων τη. Για το προβλεπόμενο μέλλον, το αμερικανικό ναυτικό με του συμμάχου αυτού θα επικρατεί σε όλη την περιοχή, ενώ η Κίνα θα προσπαθεί να προωθεί διάφορες ε, θέσεις και άλλες χώρες, θα κάνει κινήσεις στην περιοχή προσπαθώντας να δημιουργήσει ουδέτερες ζώνες στην περιοχή και να ανακτήσει ε, μια πρωτοβουλία στη Δύση μέσω του προγράμματος OBOR. Οι χώρε του ΑΣΕΑΝ θα ήθελαν μια ειρηνική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και να μπορούν να συνεργάζονται και με τις δύο χώρες χωρίς να πρέπει να κάνουν κάποια επιλογή. Η Asia προωθεί την ιδιαιτερότητά της, δηλαδή αναπτύσσει ε, σχέσεις με μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ινδία και θα μπορούσε ίσως να αυξήσει την παρουσία, της, ε, παρουσία των ΙΠΑ στην, στην Άζιαν διατηρώντας η Άσαν την ουδετερότητα και έχουν επικριθεί προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να αναπτύξουν συνεργασία με κάποιες χώρες της ΑΖΕΑΝ, διότι ε, έχουν επικριθεί, διότι έτσι αποδυναμώνουν την περιφερειακή συγκέντρωση. Είναι πολύ νωρίς τώρα να έχουμε σαφές όραμα όσον αφορά την πολιτική που θα ακολουθήσει ο πρόεδρος Τρόμπ για την περιοχή, διότι έχει κάνει διάφορες αμφίσιμες δηλώσεις που είναι αντι, αντικρουόμενες. Τώρα ερχόμαστε στο όμπορ την πρωτοβουλία Ομπόρ. Το 2013 ο πρόεδρος Τζι Jinping ανακοίνωσε ότι δημιουργεί την πρωτοβουλία μιας ζώνης, μια, ενός δρόμου κατά το τέλος του 2004, μιας διέλευσης. Η Κίνα δημιούργησε ε, μια υποδομή, ε, ασιατική υποδομή χρηματοδότησης, την Ασιατική Τράπεζα ε, Χρηματοδότησης και το Ταμείο για το Δρόμο του Μεταξιού για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει ασιατικά αναπτυξιακά προγράμματα. Για πολλούς αναλυτές η νέα στρατηγική για το δρόμο του μεταξύ στρατηγική έχει εμορφωθεί κατόπιν της ε, πιέσεω από τις ΗΠΑ να επαναξισορροπήσουν τι πολιτικέ. Μερικοί θεωρούν ότι πρέπει να αποφευθεί η αντιπαράθεση τελικά με τις ΗΠΑ. μπορεί να βελτιώσει την διεθνή τη εικόνα ε, η Κίνα σαν υπεύθυνη δύναμη και να ε, διαμορφωθεί σαν παγκόσμια δύναμη. Το μπορ μπορεί να γίνει μια εναλλακτική ε, λύση για διαμόρφωση διεθνούς πολιτικής και θα μπορούσε να είναι όχημα για δημιουργία μιας νέας πολιτικής και οικονομικής τάξης. Οι αντιδράσεις όσον αφορά την πρωτοβουλία Μπορ ποικίλουν από ενθουσιαστικές αντιδράσεις, κυρίως στην οικονομική, στον οικονομικό τομέα, μέχρι μεγάλη θετικότητα και αμφισβήτηση. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ε, έχει επιλεκτική αντίδραση. Κάποιοι αξιωματούχοι, λίγοι, της Αμερικής, ανέφεραν ή επένεσαν τη σημασία που έχει το ΟΜΠΟΡ. Απ' την άλλη πλευρά, σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς, όπου απαιτείται η βοήθεια της Κίνας όπως την συντήρηση της σταθερότητας και την ανάπτυξη στην Κεντρική Ασία έχει εκφράσει προσεκτικά ε, θετική στάση και συνεργάσιμη στάση. Ταυτόχρονα θεωρεί το όμπορ σαν αντίπαλο στο TPP που έχει ακυρωθεί. Και έτσι οι ΙΠΑ ασκούν ε, ανοιχτές πιέσεις στην ε, Νότια Κορέα και την Αυστραλία να μην συμμετάσχουν στα κινέζικα ταμεία. Μεταξύ των χωρών της ΑΣΕΑΝ υπάρχουν αντιδράσεις πιο ήπιες. Η Μαλαισία και η Ινδονησία έχουν υποστηρίξει την πρωτοβουλία. Το Βιετνάμ αντιθέτως έχει... είναι πολύ καχύποπτο και το Μιανμάρ που υπέγραψε μια συμφωνία με την Κίνα να αναπτύξει σιδηροδρομική σύνδεση ακύρωσε το όλο έργο. Η Ινδία παραμένει καχύποπτη και επανειλημμένα εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την αυξανόμενη στρατηγική και οικονομική παρουσία της Κίνας η Ινδία θεωρεί και τη ζώνη και τον δρόμο ως συνεχιζόμενη προσπάθεια περικύκλωσης και θεωρεί τη στρατηγική ως πρωτοβουλία που ανταγωνίζεται την πολιτική της στην Νότια Ασία. Ε, προβλήματα και διενέξεις λόγω συνόρων δεν έχουν επιληθεί και παραμένουν ε, ως προϋπόθεση για περαιτέρω συνεργασία με την Κίνα. Στη Σρι Λάνκα ανεστάλλει το κινέζικο πρόγραμμα για τα λιμάνια. Στην Αυστραλία η Κίνα επικρίθηκε γιατί χρησιμοποίησε τα τεράστια κεφάλαιά της για να κυριαρχήσει σε μικρότερες οικονομίες μέσα από μακροπρόθεσμο έλεγχο υποδομών, φυσικών πόρων και γης και προσφέροντας ε, λιγό, ε, ε, ε, όρους για δάνεια για υποδομές. Παρά την ε, οικονομική φύση όπως ισχυρίζονται της ατζέντα Obor, οι επικριτές θεωρούν ότι η πρωτοβουλία είναι και στρατηγικό πρόγραμμα. Έχει επανειλημμένα σημειωθεί στην Κίνα ότι το ομπόρ ε, θεωρείται και ως μηχανισμός περιφερειακής ασφάλειας με, ισχυρά, μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με το μελλοντικό ρόλο του στρατού ε, για την προστασία των εγκαταστάσεων ομπόρ της Κίνας στο εξωτερικό. Το 2013 οι Φιλιππίνες άρχισαν διαδικασίες διαιτησίας κατά της Κίνας. Ε, η Κίνα αντέδρασε απορρίπτοντας την ε, διαιτησία και επέστρεψε την κοινοποίηση και τον, ε, τη δήλωση διεκδικήσεων στις Φιλιππίνες. Το μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο από, έλαβε απόφαση ή για την Κίνα ήταν μεγάλο πλήγμα η απόφαση του δικαστηρίου ε, ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική της Κίνας. Η απόφαση είναι απαράδεκτη για το καθεστώς και θέτει ε, κάτω από ισχυρέ πιέσει στην κινέζικη κυβέρνηση για να αντιδράσει και να σώσει τα προσχήματα. Δεν εκπλήσει το γεγονό ότι το Πεκίνο απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου. Ο πρόεδρο ε, Τζιν Πίνγκ είπε ότι η δαφική κυριαρχία και τα δικαιώματα στη θάλασσα της Κίνας δεν θα επηρεαστούν από την απόφαση και είπε ότι η Κίνα όμω θέλει να επιλύσει τι διαφορέ με του γείτονε. Η ε, χώρες ΑΖΕΑΝ ε, κράτησαν χαμηλό προφίλ, ε, απέφυγαν στη, να αναφέρουν την απόφαση στην κοινή δήλωση του Βιεντιάνε τον περασμένο Ιούλιο του 2016 δηλαδή. Τώρα, ποιο είναι το follow-up, τι συνέχεια θα δοθεί. Πέρσι τον Οκτώβριο ο πρόεδρος των Φιλιππίνων ε, πήγε στο Πεκίνο και είπε στους ε, Κινέζους ότι θέλει να φιλία και όχι πόλεμο. Ο κύριος Ντουτέρτε ανακοίνωσε ότι θα ε, μείωνε τη στρατιωτική του συνεργασία με την Ουάσιγκτον και οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να ξαναρχίσουν απευθεία συνομιλίες για το πρόβλημα της Νότιας Συνικής Θάλασσας και είπαν ότι ε, θα, έχουν και, θα, δημιουργήσουν και μια κοινή επιτροπή ακτοφυλακής. Η Κίνα είπε ότι θα βοηθήσει με την υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση των ψαριών. Στις επενδύσεις ε, είπε ότι θα χρηματοδοτήσει την, ε, τις υποδομές. Ήρε το εμπάργο για τις εισαγωγές τροπικών φρούτων. Είπε ότι θα ενθαρρύνει τον τουρισμό στις Φιλιππίνες ο κύριος Ντουτέρτε είπε ότι δεν θα θέσει θέμα συνεκμετάλλευσης με την Κίνα ε, στη νότια συνική θάλασσα ε, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο πρόεδρος Ντουτέρτε ζήτησε από τους Κινέζους να βοηθήσουν τις Φιλιππίνες να καταπολεμήσουν τις ε, ένοπλες ληστείες και την τρομοκρατία στη θάλασσα Σούλου και πρότεινε να κηρύξει απαγόρευση της αλληλείας στις βραχονισίδες Κάρμπορο η οι αυξανόμενες θαλάσσιες μεταφορές στην Νοτιοσυνική θάλασσα, η στρατηγική σημασία ε, για την οικονομία της Κίνας, της περιοχής αυτής, ε, νομιμοποιούν την Κίνα να προσέξει ιδιαίτερα αυτή την περιοχή. Η Κίνα είναι κράτος με πυρηνικά όπλα. Μία από τις προτεραιότητες της Κίνας είναι να ε, έχει πυρηνική αποτροπή, συγκεκριμένα δηλαδή ε, ε, υποβρύχια στρατηγικών βαλιστικών πυράβλων. Η νότια συνική θάλασσα θα πρέπει να είναι ασφαλή για την Κίνα για την κυκλοφορία αυτών των υποβρυχίων. Ε, και η Κίνα προσπαθεί να αποκτήσει έλεγχο στη θάλασσα στα ύδατα αυτά, δηλαδή για να αντιμετωπίσει την παρακολούθηση από την πλευρά των ΗΠΑ. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μείζον παίκτη στο παγκόσμιο εμπόριο και ε, ε, εξαρτάται πολύ από τις ε, θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών στον Ινδικό και στην Κυσινική θάλασσα. Ε, τα βασικά συμφέροντα της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή Ασίας ειρηνικού συμπεριλαμβάνουν την ελεύθερη διακίνηση και ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων. Το μεγάλο, μεγάλος κίνδυνος είναι η αντιπαλότητα στις περιοχές αυτές να επηρεάσει την κατάσταση αποσταθεροποιητικά και στον Ινδικό και στην Νότια Συνική Θάλασσα και να αποσταθεροποιήσει έτσι και περιοχές στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας είναι κυρίως οικονομικές και εμπορικές. Οι οικονομικές ανταλλαγές είναι σημαντικές και με τις χώρες ΑΖΕΑΝ, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία και όλες περνούν από τις ε, θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα υπέγραψαν Συμφωνία Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας το 1985 που αποτελείται από τρεις πυλώνες ε, ε, για το διάλογο ε, πολιτικές ανταλλαγές οικονομικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές. Το 2013 μια στρατηγική συνεργασία εγκρίθηκε Κίνα Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 που δεν συμπεριλάμβανε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Η Κίνα είναι ο πρώτος προμηθευτής Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης ο πρώτος ε, σε παροχές για την Κίνα το 2015. Το εμπορικό ε, έλλειμμα με την Κίνα έφτασε 180 δις ευρώ. Οι ε, πολλές, πολλές διαφωνίες και διαφορές στο εμπόριο υπάρχουν, αλλά είναι περισσότεροι οικονομικοί δεσμοί τώρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. τώρα η απόφαση του Τραμπ κατά τη συμφωνία TPP μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρία για μια νέα προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Ε, για την ΑΖΕΑΝ, η κυρία Μαγκερίνη δήλωσε ότι η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΑΖΕΑΝ είναι πολύ μεγάλη σημασίας. Για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες το 2014 ε, μπήκαν στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής ε, θέματα ασφάλειας τον Ιούλιο του 2016 ε, αποφασίστηκε ε, να αρχίσει η διαδικασία για μια στρατηγική εταιρική σχέση ΑΖΕΑΝ-Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξηθεί η συνεργασία. Ε, υπάρχουν πιθανόν κάποιοι τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ομπόρ της Κίνας ή με τα προγράμματα άλλων χωρών, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τις δικές της αξίες και το όραμα σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις. Αν και οι Κινέζοι ηγέτες δηλώνουν ότι η Ασία είναι ανοιχτή στον κόσμο, επαναλαμβανόμενες θέσεις όπως η Ασία για τους Ασιάτες και ε, η κοινότητα ε, ε, μιας ενιαίας μοίρας θεωρούνται μια, ένα χλωμό αντίγραφο του δόγματος Μονρό των Ηνωμένων Πολιτειών για την Αμερική, Βόρεια και Νότια όπως και παρόμοια ε, προγράμματα της Ιαπωνίας. Ε, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν καθιερώσει διεθνές δίκαιο και πρότυπα τα οποία διέπουν σήμερα τον κόσμο. Με την εξαίρεση και υπάρχει συνεργασία ε, στην, ε, οι, Πολιτι... το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ε, έχει φύγει από την Μεσόγειο με την εξαίρεση τέσσερα αντιτορπιλικά στην Ισπανία. η εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ θα μπορούσε να είναι ανησυχητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πολλών δηλώσεων σχετικά με τον απομονωτισμό των ΗΠΑ εδώ. Ε, από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τον επεκτατισμό της Κίνας συμπεριλαμβάνοντας ε, τα προβλήματα διεθνούς δικαίου. Από την άλλη πλευρά η στρατηγική αντιπαλότητα μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας θα μπορούσε να συγκλονίσει την παγκόσμια οικονομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, διαλέξει ε, σε, με ποιο το μέρος θα πάει αν υπάρξει τέτοια διένεξη. Ε, σχετικά με το ούγκλος η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, ε, σήκωσε, δεν, ακούστηκε με τρόπο ηχηρό σχετικά με τη διένεξη για τη Συνική Θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχθεί την στάση της Κίνας βέβαια και θα πρέπει να ε, υπερασπιστεί την απόφαση του δικαστηρίου. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για συζήτηση μεταξύ των διεκδικούντων. Για να επιληθεί το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρήσει το στρατηγικό ενδιαφέρον της Κίνας ε, ε, για την ναυτική βάση Γιουλίν στην Χαϊνάν θα πρέπει να το λάβει υπόψη αυτό δηλαδή και να ε, συμβουλεύσει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στο, για τη Νότια Συνική Θάλασσα. Ακόμα και αν αυτό δεν συνάδει με τις απόψεις των ΗΠΑ. Τώρα, οι πολιτικές επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η, η προσέγγιση είναι ήπια ε, η εστίαση είναι το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρείται ισχυρός ε, ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας. Ε, οπότε θα μπορούσε να ε, ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός μηχανισμού διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να μετριάσει τα προβλήματα. Οι πολιτικές επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να είναι οι εξή. Πρώτον, σύμφωνα με την παγκόσμια, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη δράση θα είναι να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη ένωση που θα εδράζεται σε κοινέ αξίες, αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να συζητεί επίση όρι με τι μεγάλε δυνάμει. Δεύτερον, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε ε, προήγαγε το διεθνές δίκαιο ως βάση για την θαλάσσια διακυβέρνηση και δεν μπορεί να δεχτεί την απόρριψη από την πλευρά της Κίνας της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Ε, κατόπιν τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει για να αποφύγει αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και είπα στην νότια Συνική θάλασσα, πράγμα που θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις θαλάσσιες μεταφορές και στο παγκόσμιο εμπόριο. Ε, η ανάπτυξη ενός κώδικα δεοντολογίδας στην νότια Συνική θάλασσα θα μπορούσε να επιχειρηθεί με διμερείς και πολυμερείς συζητήσεις. Αυτό είναι καλό για να βρεθεί συμφωνία ε, σχετικά με τις ΑΟΖ, την αλληλεία, περιβαλλοντικούς κανόνες, την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή ε, και λαμβάνοντας υπόψη επίσης, να λάβει υπόψη επίσης και την στρατηγική πυρηνική αποτροπή της Κίνας. Η πρόταση της, ε, της ολοκληρωμένης ε, θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης ως βάση για τη συζήτηση θα μπορούσε να βοηθήσει. Όπως ανέλησε η ύπατη εκπρόσωπος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντατικοποιήσει τη σχέση με την ΑΖΕΑΝ, αυξάνοντας την παρουσία της και ε, διευκολύνοντας την πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην ΑΖΕΑΝ. Η ευρωπαϊκή πολιτική προς την ΑΖΕΑΝ ανταγωνίζεται το ε, πρόγραμμα ΟΜΠΟΡ της Κίνας. Για την ΑΖΕΑΝ αυτή η αυξανόμενη δεσμή με άλλες χώρες ε, είναι ευπρόσδεκτη και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Ε, προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα να μην υπάρχει αποκλειστική ή υπερβολική εξάρτηση από την Κίνα. Η εξέλιξη της στρατηγικής της Κίνας και η κατάσταση στην Ανατολική και Νότια Συνική θάλασσα ε, απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Αυτό απαιτεί συλλογή πληροφοριών από τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών για καλύτερη ε, ενημέρωση και λήψη αποφάσεων. Τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνάδουν πάντοτε με εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελείται αν υιοθετήσει πιο ανεξάρτητη θέση σε θέματα ασφάλειας σε σχέση με την Ασία. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει επίσης να ε, λάβουν υπόψη του ότι σχέση με τις ΗΠΑ έχουν αλλάξει και θα συνεχίσουν να εξελίσσονται. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρέχει λιγότερη υποστήριξη και θα αποστασιοποιηθεί από, από τους Ευρωπαίους ε, συμμάχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών, να αυξήσει τις αμυντικές προσπάθειες και να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο ΝΑΤΟ. Η νέα αυτή ισορροπία από πλευρά είπα, προς την Ασία προϋποθέτει ε, ε, ότι η Ευρώπη θα αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη σταθερότητα στην άμεση ε, περιοχή της, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και την Αφρική. Όλοι οι παρατηρητές συμφωνούν ότι η επιχείρηση Αταλάντα στο κέρας της Αφρικής είχε επιτυχία. Η... Παρά τις δυσκολίες της αποστολής, η επιχείρηση Σοφία ε, έσωσε ζωές μεταναστών και βοηθεί τη Λιβιβύη. Ε, μία μόνιμη ενεργοποίηση του Euromar 4 ε, στην ε, Μεσόγειο και στη ακτή της Δυτικής Αφρικής θα μπορούσε να δώσει τα απαραίτητα μέσα για την παρουσία και επαγρύπνηση στη θάλασσα, η παρακολούθηση, εκπαίδευση, πρόληψη κρίσεων κλπ. Η επαγρύπνηση στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια. Οι ίπα αναπτύσσουν το σύστημα ΜΙΣΕ, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση το σύστημα ΣΥΣΕ, οι ε, χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν το IFC, το Information Fusion Center, Σιγκαπούρη. Η σύνδεση μεταξύ των ε, δικτύων αυτών θα βελτιώσει σημαντικά την θαλάσσια παρακολούθηση και επαγρύπνηση. Επίσης, ε, το ΟΜΠΟΡ ανοίγει ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει γεωστρατηγικές φιλοδοξίες στην Κεντρική Ασία εμβαθύνοντας τη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας μέσα από τη συνεργασία σε μη παραδοσιακούς τομείς ασφάλειας όπως ε, αποφασίστηκε το 2007 και επιβεβαιώθηκε το 2015. Αυτό ενδεχομένως θα προλιάνει το έδαφος για μια συμφιλίωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία. Μπορεί να είναι επωφελές για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει πώς οι, οι φυστάμενοι μηχανισμοί για την πολιτική της και, τη στρατηγική της θα μπορούσαν να συνδυαστούν με το ΟΜΠΟΡ. Τέλος, οι νέες πρωτοβουλίες της Κίνας θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της επιρροής της ε, στη θάλασσα και στην Ασία και την Αφρική και την Ευρώπη. Ε, μια προορατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με στενή συνεργασία με τοπικούς παίκτες και συντονισμό των δράσεων ή των προγραμμάτων με την Κίνα φαίνεται να είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων και του ρόλου της Ευρώπης. Για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματικό συμφέρον να στηρίξει την ε, στρατηγική ε, ολοκληρωμένη στρατηγική για τη θάλασσα της Αφρικής για το 2050 για να βελτιώσει ασφάλεια, να αντιμετωπίσει παράνομη μετανάστευση, πειρατεία ε, και να βελτιώσει και την οικονομία των αφρικανικών χωρών σε συντονισμό με επενδύσεις ε, της Κίνας. Ευχαριστούμε πολύ Ναύαρχε για την πληρέστατη αυτή παρουσίαση. Ακούσατε λοιπόν πάρα πολλές πτυχές της περιγραφής της κατάστασης στην Νοτιοανατολική Ασία, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες ισορροπίες. Εγώ ως τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι εκπροσωπώντας την υποεπιτροπή, το λέω ξεκάθαρα αυτό, θα έλεγα ότι υπάρχει μία παλαιομοδίτικη αντίληψη μιας ε, συμμαχίας αμυντικής, δηλαδή μας δεσμεύουν κάποιες αξίες και κάποιες νομικές υποχρεώσεις επί τη βάση πολυμερών συμφωνιών προκειμένου να αμυνθούμε κατά εξωτερικών απειλών. Βεβαίως υπάρχουν μηχανισμοί για κάτι τέτοιο. Εντός του ΝΑΤΟ υπάρχει το άρθρο 4, αλλά ίσως ό,τι αφορά στις πολιτικές αναλύσεις υποχρεούμεθα κατά κάποιον τρόπο να ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Παρότι λοιπόν υπό την έννοια της επιστημονικής ανάλυσης πρέπει να εξετάζουμε όλα τα σενάρια και όλα τα τμήματα αυτής της περίπλοκης εικόνας με δυνητικές πιθανότητες η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα είναι ότι συνδεόμαστε με, κάποια, με κάποιους εταίρους κάποιους εξωτερικούς εταίρους έτσι έχουν και τα πράγματα κατά την άποψή μου και στην περίπτωση της ε, αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας γιατί παρά τον την βαθιά εκτίμηση και σεβασμό που έχουμε για την κινέζικη κουλτούρα και τον κινέζικο λαό, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις πολιτικής ως προς το κινέζικο κράτος και τη σχέση του και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί παραδείγματι, το εμπορικό ισοζύγιο ή ισορροπία, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ημών και της Κίνας σχετίζεται με πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό της Κίνας και πολύ χαμηλότερα πρότυπα σε πολλά επίπεδα, το οποίο δημιουργεί προβλήματα και κοινωνικής ασφαλείας. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση. Η δεύτερη είναι ότι εξετάζοντας το νομικό πλαίσιο σχετικά με την μη επικύρωση της ούγκλος αφενός και των μη ευνοϊκών αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου επί της Κίνας αφετέρου, η πηγή των δύο δυναμιών δεν είναι η ίδια. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, σεβόμενος κανείς υψηλού επίπεδου κριτήρια, τα τοποθετεί αυτά στη βάση της πολιτικής του. Όταν όμως αυτό δεν επικυρώνεται, γίνεται πολύ διαφορετικό. γιατί είναι η νομική αιτιολόγηση των επιχειρήσεων, αλλά όταν δεν το επικυρώνει κανείς, η αμερικανική αδυναμία βρίσκεται, εντοπίζεται απλώς στη νομική διαφορά που έχει με τις Φιλιππίνες και την Κίνα. Δηλαδή η νομική επιχειρηματολογία δεν είναι καθόλου η ίδια. Η Κίνα δεν εκπληρώνει τις διεθνείς της νομικές υποχρεώσεις, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε εκπληρώνουν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, χωρίς όμως να έχουν επικυρώσει. Αυτό δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Είναι τελείως διαφορετικό πεδίο, θα έλεγα. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό είναι απλώς η δική μου σκέψη ο συνάδελφος, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Ναι, μετά βεβαίως, λέει η πρόεδρος. Ο κύριος Μπούχνα. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομη ερώτηση. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πρέπει να παίξουμε μεγαλύτερο ρόλο στην ε, περιοχή μας αλλά και στην περιοχή, δηλαδή και στον Ινδικό και στον κόλπο της Γουινέας. Πώς θα πρέπει να βελτιώσουμε την παρουσία μας, την επαγρύπνησή μας ως ναυτική δύναμη. Τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς. Ευχαριστώ. Yeah. Yeah you Εάν δεν ζητάει κάποιος άλλος το λόγο, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Αβαρχό για την παρουσίαση, η οποία καλύπτει ένα ευρύτατο έδαφος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συζητήσουμε όλες τις διάφορες ενδιαφέρουσες πτυχές που φύγει. Εγώ θεστιζόμουν στην νοτιοανατολική θάλασσα και ίσως και στο όμπορ. Πρώτα απ' όλα, η κινέζικη διεκδίκηση στην νότια κινέζικη θάλασσα έχει μεταβληθεί, μεταξελιχθεί συν το χρόνο. Η λεγόμενη γραμμή 9 Παύλα που αρχικά ήταν 11 παύλα μας οδηγεί στην απορία του πώς χάθηκαν δύο παύλες που σημαίνει ότι η Κίνα απόλυσε δύο παύλες προκειμένου να βοηθήσει τον Χότσι Μίνχ ε, στον πόλεμο κατά των Πολιτειών. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα πω ότι δεν πρόκειται για μια διεκδίκηση η οποία ήταν απολύτως παγιωμένη στο χρόνο. Υπήρξε και μια μελέτη αμερικανική πριν από κάποια χρόνια που έλεγε ότι οι εννέα παύλες έχουν μετακινηθεί πιο κοντά, πολύ πιο κοντά, στα σύνορα των γειτονικών χωρών. Τώρα πέρα του διατητικού πάνελ της Ούγκλος πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κατά την οποία η Κίνα μπορεί να υποστηρίξει τις διεκδικήσεις με τρόπο που δεν μπορεί καμία άλλη χώρα στην περιοχή. Και παρότι αξίζει να επιμένουμε στο διεθνές δίκαιο, που το τηρούμε όλοι και που όλοι προσυπογράφουμε σε αυτό, πρακτικώς μιλώντας, η πολιτική μας δεν μπορεί να κατευθυνθεί προς τη βοήθεια οποιασδήποτε άλλης διεκδίκησης από την Κινέζικη προς την εκπλήρωση δηλαδή της φιλοδοξίας της. Θα πρέπει να συνεισφέρουμε στο μέτρο του δυνατού να διατηρήσουμε και να διατηρούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Διότι έχουμε συμφέρον να το κάνουμε αυτό. Υπό την έννοια αυτή έχουμε και εμείς, όχι διεκδίκηση, αλλά εν πάση περιπτώσει συμμετοχή στο όλο σύστημα. Η κατάσταση σταδιακά έχει οδηγήσει σε μια πιο ισχυρή θέση της Κίνας και σε μια μεγαλύτερη δυνατότητα της Κίνας να επιβάλλει τις απόψεις της. Αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια της όλης κατάστασης, αλλά και στην ασφάλεια της Ταϊβάν, το οποίο δεν ανεφέρθη, αν δεν κάνω λάθος, από τον Άβαρχο. Που όμως και αυτό εμπίπτει στη συνολικότερη εικόνα. Εγώ δεν θα ήμουν υπέρ μιας ερμηνεία που θα έλεγε ότι αυτή εδώ είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις μεταξύ της Κίνας και των γειτόνων της. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ως ε, παγκόσμια δύναμη που είναι δίνει μεγάλη σημασία στην ελευθερία των ανοιχτών θαλασσών και έχει τοποθετηθεί σταθερά όχι στο ποια βραχονισίδα ανήκει σε ποιον, αλλά στην εφαρμογή, στην επιβολή του διεθνούς δικαίου. Και θα ενίσχυε τη θέση των ΗΠΑ να ξεπεράσουν την ανόητη άρνηση της γερουσίας να επικυρώσει την Ούγκλος. Όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών έχουν ζητήσει ξανά και ξανά ανεξαρτήτως του κόμματος το οποίο ανήκαν από τη Γερουσία να επικυρώσει. Και δείχνει χαμηλή αξιοπιστία η θέση των ΗΠΑ να προσπαθούν να επιβάλλουν την ούγκλος την οποία δεν έχουν οι ίδιοι επικυρώσει. Σε αυτό το πεδίο δεν βλέπω κανένα ρόλο για εμάς και θα συνιστούσα να μην ακολουθήσουμε την επιλογή υπαριθμών 2 να βοηθήσουμε στην επίλυση της αντιπαράθεσης στην νότια Κινέζικη θάλασσα. Δεν είμαστε καν ικανοί να διαδραματίσουμε ενεργή ρόλο εκεί. και κανείς από τους συμμετέχοντες εντόπιους δεν θα μας καλωσόριζε. Μπορούμε να βοηθήσουμε τη σταθερότητα ακολουθώντας μία διτή προσέγγιση αφενός να επιμείνουμε υπομονετικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Εθνούς Δικαίου και αφετέρου να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και τη στρατηγική μας ε, εταιρική σχέση με την κοινότητα ΑΣΕΑΝ, όπου η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να αφιερώσει περισσότερη προσπάθεια ώστε οι χώρες αυτές να μείνουν μαζί και να αποφύγουν τις φυγόκεντρες δυνάμεις που προσπαθούν να διασπάσουν το σύνολο αυτό. και για μια οποιαδήποτε διπεριφερειακή FTA μεταξύ της ΑΣΕΑΝ και η μόνη άλλων, κάτι τέτοιο θα είχε μια γεωπολιτική αξία, πιστεύω, πέραν της καθαρά οικονομικής ή εμπορικής της αξίας. Τελευταία παρατήρηση για το όμπορ. Το όμπορ είναι κάτι περισσότερο από στρατηγική, θα έλεγα. Είναι ένα σχέδιο μιας νέας παγκόσμιας τάξης που οργανώνεται σύμφωνα με το παράδειγμα Hub and και Spokes. Αυτό είναι απολύτως αντίθετο προς την αρχή του, της πολυμερούς προσέγγισης προς την οποία, την οποία μάλλον έχουμε σεβαστεί πάντοτε. Η Κίνα είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς ότι έχει προσκαλέσει τους πάντες να συμμετάσχουν στο όμπορ. Η μόνη χώρα που η απουσία της είναι σαφής στην πρόσκληση αυτή παρότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις μελλοντικέ διόδους του όμπορ είναι ακριβώς οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αναπόφευκτα λοιπόν θα πρέπει με μια πολύ πρακτική προσέγγιση να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που υφίστανται στο πλαίσιο όμπορ Πρέπει να αποφύγουμε να αγνοήσουμε το όλο πλάνο, το όλο πλαίσιο. Πρέπει μάλλον να καταλάβουμε πού θα οδηγούσε και δεν είμαι βέβαιος ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν πάντοτε επιδείξει μια τέτοια πλήρη κατανόηση. Τίνω να συμφωνήσω μαζί σας με την τελευταία σας παρατήρηση, λέει η Πρόεδρος. Και επί τη βάση της πολιτικής των μεμονωμένων κρατών μελών. Είναι τελείως διαφορετικό. Νομίζω όμως, Ναύαρχε, ότι ήρθε η ώρα για το δεύτερο γύρο των παρατηρήσεών σας και θα σας ζητούσα μια διευκρίνηση ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος της ύπαρξης της φράσης για την οδό προς τη συμφιλίωση με τη Ρωσία, λέει η πρόεδρος Φωτίγκα. Γιατί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην περιοχή μου, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αυτό είναι ένα προφανές ζήτημα. Παρακαλώ. Περισσότερη σαφήνεια. Θα μιλήσω γαλλικά για να είμαι πιο σαφής. Πρώτα απ' όλα το θέμα που αφορά το θαλάσσιο τομέα. Διαπιστώνω ότι κανείς ε, δεν είναι στη Μεσόγειο. Κανείς, τι εννοώ, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι έχουν εγκατασταθεί και παρά την επιχείρηση Σοφία η Ευρώπη είναι απούσα. Δεν είναι παρούσα, δεν είναι ορατή. Είναι αποδεκτό αυτό. Είναι αποδεκτό σε αυτή τη ζώνη που έχει προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα να μην έχουμε την ευρωπαϊκή σημαία μονίμως ε, ε, παρούσα στη θάλασσα για μένα όχι. Για μένα που είμαι και θαλασσινός όχι. Είμαστε παρόντες με την Αταλάντα στον Ειδικό ωκεανό, πολύ καλά. Έχει γίνει εξωσημείωτη δουλειά. Εκτι... Την εκτιμούν. Έχει αρχίσει να νοθώνει τη Σομαλία. Η πειρατεία έχει εξαλειφθεί ουσιαστικά. Υπάρχουν και άλλες περιοχές ε, που επηρεάζουν τα μέσα συμφέροντά μας. Και το να έχουμε μια ευρωπαϊκή θαλάσσια δύναμη στον κόλπο της Γουινέας όπου έχουμε συμφέροντα όσον αφορά το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, οικονομικά συμφέροντα. Θέλουμε να αναπτύξουμε εμπόριο με την Αφρική, μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την Αφρική τόσο σε αυτή η μετανάστευση η οποία μας ρηπαίνει, λομιλητής και δημιουργεί πραγματικές δυσκολίες στην Ευρώπη ε, εξακολουθεί να εφίσταται. Έχουμε κάθε συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα και μπορεί ε, η θαλάσσια δύναμη να συμβάλλει ποικιλοτρόπω, αυξάνοντα την ασφάλεια και σταδιακά μπορούμε να δώσουμε ε, τον έλεγχο στις αφρικανικές χώρες, στις θαλάσσιες δυνάμεις, στις ναυτικές δυνάμεις των αφρικανικών χωρών. λοιπόν, απευθύνω μια έκκληση να έχουμε μια παρουσία ορατή ευρωπαϊκών δυνάμεων ε, στα, στη δική μας ε, άμεση περιοχή και γειτονιά. Όταν έκανα, συμμετείχα στο επιτελείο στη Γαλλία, προσπάθησα να δημιουργήσω αυτή τη διασύνδεση, αυτή τη σχέση, να δημιουργήσω μια πολυεθνική δύναμη στον κόλπο της Γουινέας. Είμαστε εκεί από το 1996 χωρίς να είμαστε πραγματικά επιτυχείς. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει σταδιακά να φτάσουμε στο να έχουμε μια τέτοια παρουσία ε, πολυσυμμετοχική, ε, ευρωπαϊκή, ορατή. Αυτή την απάντηση μπορώ να δώσω στην τεθήσα ερώτηση. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες ερωτήσεις, που είναι πολύ σημαντικές, αφορούν σημαντικότητα ζητήματα, να πω πώς προσέγγισα για να αναλύσω το θέμα που μου ανετέθη. Έχω επίγνωση ότι ξεπέρασα το απλό πρόβλημα της ελευθερίας των θαλασσών στην ανάλυση μου, διότι για μένα όλα είναι αλληλένδετα. Και αυτό που συμβαίνει όταν συζητούμε τις γραμμές επικοινωνιών, θαλασσίων επικοινωνιών, είναι μιλάμε ε, για τα κινέζικα λιμάνια και φτάνουμε σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Πρέπει να εξετάσουμε μια ολόκληρη λυσίδα με ολόκληρη ζώνη να δούμε πού βρίσκονται οι κίνδυνοι και πού βρίσκονται τα αδύνατα σημεία. Η Ευρώπη περισσότερο από άλλη χώρα έχει συμφέρον να μην υπάρξει σύγκρουση στην νοτιοανατολική συνική θάλασσα. Αν μιλάμε για αυτή την βασική υπόθεση λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να αποφευθεί μια τέτοια σύγκρουση εκεί και ε, διατείνομαι ότι υπάρχουν εργαλεία που κανένα στον κόσμο δεν έχει αναπτύξει σήμερα και κυρίως η, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική η οποία είναι αξιοσημείωτη και που θα ήθελα και θα ευχόμουν ε, να είχε δημιουργηθεί το 2007, δημιουργήθηκε το 2007 και θα πρέπει να επαναπροωθηθεί τώρα διότι είναι ακρογωνίως λήθος ε, μια σημαντικότατη βάση για τις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και που συνάδει πλήρως με το όραμα προστασίας του περιβάλλοντος που έχουμε, της προστασίας του πλανήτη μας και είναι ένας τρόπος να διευθυντήσουμε τις διαφορές όσον αφορά τον τομέα των θαλασσών. Λοιπόν, μας περιβάλλει αυτός ο θαλάσσιος χώρος. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μην προτείνουμε μια τέτοια λύση, αυτή που βρήκαμε εμείς στις χώρες ε, που προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο με μια χώρα που προσπαθεί να εφαρμόσει την αρχή του ε, τετελεσμένου γεγονότος που οδηγεί σε αδιέξοδο κατά την άποψή μου και δημιουργεί κινδύνους και μπορεί να εμποδίσει μακροπρόθεσμα και την ανάπτυξη της χώρας της μεγάλης αυτής μπορούμε να παίξουμε το δόλο της ε, δύναμης που δεν ε, ε, βλάπτει κανένας προσφέροντας εφικτές λύσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε να επιληθεί αυτή η διαφορά στη θάλασσα της Κίνας και πιστεύω ότι η πρωτοβουλία του Προέδρου των Φιλιππίνων μπορεί να είναι σωστή προσέγγιση. Θα πρέπει και αυτή όμως να προσχωρήσει αυτό το όραμα όλες οι χώρες, η Μαλαισία, το Βιετνάμ, όλες οι χώρες που ενδιαφέρονται να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα και έχουν διεκδικήσεις. Ε, είναι δύσκολο, αλλά απαιτεί μεγαλύτερη παρουσία μας στα διάφορα βήματα, στους διάφορους χώρους και να πιστεύουμε σε αυτό που προτείνουμε και σε αυτό που έχουμε υλοποιήσει. Ε, και εκεί λέω και εγώ ότι υπάρχει ανάγκη να έχουμε ισχυρότερη Ευρώπη πιο σίγουροι για τις αξίες της. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολιτικοί στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με δυστυχώς ε, κίνδυνο να καταρρεύσει ένα οικοδόμημα που κατασκευάστηκε υπομονετικά και δυστυχώς καταραίει. Αν δεν είμαστε ισχυροί εσωτερικά αν δεν έχουμε παγιώσει τις δομές μας, δεν θα έχουμε βάρος έναντι χωρών που είναι τόσο ισχυρές όπως είναι η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό ήθελα να πω. Η ΑΖΕΑΝ είναι μια δομή, όχι τόσο περίπλοκη ως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντικατοπτρίζει αυτά που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε εμείς. Είναι ένας εταίρος για το μέλλον. Μας χρειάζεται και μπορούμε αμοιβαίως να ισχυροποιηθούμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα στην περιοχή. Όχι μόνο στραφούμε κατά τον ΙΠΑ ή της Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική που πρέπει να προωθηθεί και που πιστεύω ότι είναι μια πολιτική να ανοίξει το δρόμο προς λύσεις. Επέμεινα λέγοντας ότι πέρα από το σεβασμό της ελευθερίας των θαλασσών και του σεβασμού των κανόνων τη συμβάσεω του Montego Bay, του UNCLOS, υπάρχει κάτι στο οποίο θα υποχωρήσει ποτέ η Κινέζοι. Η ασφάλεια των στρατηγικών του πυρηνικών όπλων, των, των πυρηνικών του δυνάμεων, όπως και στη χώρα μου, το γνωρίζετε γίνεται στη χώρα μου, είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Άρα θα πρέπει να συζητηθεί. Έχει δικαίωμα να προστατεύσει τα πυρηνικά της υποβρύχια που εξασφαλίζουν την άμυνά της. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και πρέπει να δούμε πώς αυτό μπορεί να ενταχθεί και να συμπεριφθεί στις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν με την Κίνα ε, στο μέλλον. Όσον αφορά το το σχέδιο BOR συνδέεται με όλα αυτά τα ζητήματα ε, ε, έχουμε τη χερσαία προσέγγιση έχουμε και τη θαλάσσια ε, προσέγγιση. Πρέπει να δούμε σχετίζεται τα, τα συμφέροντα των θαλασσών με τα συμφέροντα της χερσαίας επικράτειας. Πρέπει να συζητήσουμε τα ζητήματα αν θέλουμε να υπάρχουν εξελίξεις. Η Ρωσία είναι μια χώρα που το θέλουμε είτε όχι, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί μπορούμε να προσπαθήσουμε ε, να εφαρμόσουμε προληπτικά μέτρα αντί της Ρωσίας. Θέλουμε να στραφεί η Ρωσία προς την Κίνα. Μας συμφέρει να δημιουργηθεί ένα μπλοκ που θα προσπαθήσει να εφαρμόσει παγκόσμια διακυβέρνηση από αυτή που έχουμε δημιουργήσει με διαφορετικούς νόμους και προδιαγραφές κλπ. κλπ. Τίθενται τέτοια ερωτήματα. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικότατα. Αυτά ήθελα να θέσω επιτάπητος, λέγοντας ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα καταλήβηματα. Μελετώ και τι γίνεται και στην Αρκτική. Είναι μια περιοχή που για την ώρα η Αρκτική δεν έχει πληγεί από τη γνωστή προβληματική Κρυμαία, Ουκρανία κλπ. Εξακολουθούν οι σχέσεις να εφίστανται στην Αρκτική και είναι καλό η Νορβηγία και η Ρωσία έχουν, συνεχίζουν τις ασκήσεις έρευνας και διάσωσης και καταπολέμησης της ρήπανσης. Αυτό καταδεικνύει ότι πέρα από τις συμβατότητες και τα σφάλματα που διαπράττει ο καθής, μπορούμε κάπου να βρούμε που υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων και από εκεί που αυτή η σύμπτωση και η προσπάθεια για σύμπτωση συμφερόντων πιο σημαντική από πάγιες και άκαμπτες θέσεις. Και κάτι άλλο. Θα ήθελα και οι Αμερικανοί υπογράψουν τη σύμβαση. Δεν μας διαφεύγει ότι το μόνιμο δικαστήριο διατησίας άρχισε να ακούει τα αιτήματα του, τα αιτήματα του Βιετνάμ και άλλων χωρών να είναι παρατηρητές. Ζήτησαν και αυτοί και οι Αμερικανοί να είναι παρατηρητές, αλλά επειδή δεν υπέγραψαν τη σύμβαση, τους το αρνήθηκαν. Είναι όριο. Άμα δεν έχετε υπογράψει, τους είπαν, δεν μπορείτε να είσαστε παρατηρητές να ακούτε τις συζητήσεις. Άρα προς όφελός τους θα ήταν και αυτοί να υπογράψουν την, τη σύμβαση. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλατε κι εσείς να λάβετε το λόγο κύριε Βιτικόφερ. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσω κάποιες παρατηρήσεις του Αντιναβάρχου. Ε, παρουσιάσατε κάποιες ε, θέσεις ε, λίγο οξίες. Νομίζω ότι είναι υπερβολική η θέση σας σε σχέση με Ρωσία-Κίνα. Είπατε ότι η ΑΣΕΑΝ επίσης ε, ε, είναι ένα αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία χώρα δεν θα ε, συμφωνήσει. Επίσης είναι λίγο παράλογο ή γκροτέσκο να θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει 100% ε, διαφοροποίηση από τις ΙΠΑ. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια βάση συνεννόησης Ένωσης Ρωσίας και ε, θα ναι, και για την εισβολή στην Κρυμαία και την Ανατολική Ουκρανία είπατε όλοι κάνουν λάθη. Υπερβολικό. Αυτό όμως το οποίο απορρίπτω 100% είναι αυτό που λέτε ε, ε, για την για την ε, μετανάστευση η οποία ε, μας κατατρέχει. Αυτό ε, είναι μια δήλωση που φτάσετε κατά των ανθρώπων και δεν, μπορώ να το, δεν είναι μια φράση που μπορούμε να δεχτούμε. Άλλος κανείς ζητεί το λόγο. Όχι, θα απαντήσει ο κύριος Εμπράρ. Έχετε το λόγο. Ε, λυπούμε που έγινε τέτοια ερμηνεία της παρατήρησής μου. Δεν ήταν καθόλου η πρόθεσή μου αυτή. Να αποκλείσω δηλαδή το οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω ότι είμαι υπέρ της εξέβρεσης λύσεων στις τάσεις που έχουν αναπτυχθεί, στις πιέσεις και στις αντιπαραθέσεις. Μάλλον εκφράστηκα με λανθασμένο τρόπο, αλλά καθόλου δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Καθόλου. Μάλιστα. Ναύαρχε, ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ήθελα να πω ότι προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την υποεπιτροπή όσο πληρέστερη μπορούσαμε με εμπειρογνωμοσύνη και προσπαθώντας να έχουμε μια επιστημονική προσέγγιση. Επομένως το προηγούμενο σχόλιο μου ότι προσπαθούμε να εκτιμήσουμε διάφορα σενάρια αντικειμενικά και από κάθε οπτική δυνατή γωνία ακριβώς αυτό εννοούσε ότι προσπαθούμε να δείξουμε διάφορες επιστημονικές αναλύσεις, διάφορες απόψεις και εγώ προσωπικά έχω τις δικές μου απόψεις, αρκετά έντονες ενδεχομένως, αλλά αντιλαμβάνομαι απολύτως την ανάγκη της διαφορετικότητας των απόψεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. σχετικά με, τις, με τα διάφορα επίπεδα στα οποία μπορεί να καταλάβει κανείς αυτές τις απόψεις. Εμείς πρέπει να λάβουμε αποφάσεις επί τη βάση των καλύτερων αναλύσεων που έχουμε και συνήθως το κάνουμε αυτό στο Κοινοβούλιο μέσω ψηφοφορίας. Υπάρχουν πολλές και διάφορες εκθέσεις και ψηφίσματα τα οποία συνθέτουν όλα μαζί την επίσημη φωνή μας, θέση μας. Αλλά είμαστε ένα βήμα συζήτησης και μελέτης. Σας ευχαριστώ πάντως Ναύαρχε για την μελέτη αυτή παρά την ποικιλομορφία των απόψεων που εκφράζουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. short break for Ένα σύντομο διάλειμμα ε, για πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Καθίστε παρακαλώ. Φτάσαμε στο τελευταίο σημείο της ε, σημερινής ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την παρουσίαση μιας μελέτης που ζήτησε η ΣΤΟΑ και συντάχθηκε και παρουσιάστηκε στη ΣΕΝΤ και τώρα έχω την χαρά να καλωσορίσω τον συντάκτη της μελέτης, τον κύριο Παναγιώτη Τριμίντζιο, ο οποίος εκπροσωπεί το πρόγραμμα των τριών C, το C3, στην ΕΝΙΣΑ. Το θέμα είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο, στη κοινή πολιτική ασφάλειας άμυνας ε, έγινε όπως είπα ε, μια συνεργασία Ε, η μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, είναι ανοιχτή σε συνεργασίες και με το ΝΑΤΟ. Ο κύριος Τριμίτζιος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να με ακούτε όλοι. Να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην Επιτροπή. Την επόμενη ώρα θα σας παρουσιάσω με τα προσωρινά αποτελέσματα της μελέτης για τα στοιχεία του κυβερνοχώρου στα πλαίσια της ε, ασφάλειας, κοινής ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και στα πλαίσια της μελέτης θα προσπαθήσουμε να δούμε προκλήσεις και κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες πολιτικές επιλογές που μπορούμε να προτείνουμε. Η παρουσίαση τώρα με τον ε, συνάδελφο Γιώργο Χατζηχρήστο θα σας ε, κάνουμε την ανασκόπηση, το ιστορικό της μελέτης, πώς δηλαδή έφτασε να αναλάβουμε τη μελέτη, πώς μας ανατέθηκε, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα, το καθεστώς, το, πλαίσιο της μελέτης. Μετά θα δούμε πιο πολύ τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Θα σας μιλήσουμε για τις προκλήσεις, προκλήσεις πολιτικής στον τομέα του κυβερνοχώρου και της κοινή πολιτικής ασφάλειας άμυνας, ε, προκλήσεις και ε, οικοδόμηση ικανοτήτων ε, είναι πιο γενικά ε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας ε, άμυνας και τέλος θα μιλήσουμε για τον κυβερνοχώρο και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Τέλος θα παρουσιάσουμε κάποιες ε, εναλλακτικές, κάποιες επιλογές πολιτικής. Το έργο αυτό συνεχίζεται. Αυτά που θα πούμε στηρίζονται στην ενδιάμεση, στα ενδιάμεσα αποτελέσματα της μελέτης, ε, θα οριστικοποιηθεί σε λίγες εβδομάδες. Προχωρήσαμε αρκετά μετά την ε, προσωρινή έκθεση. Η παρουσίαση που βλέπετε σήμερα είναι πιο κοντά προς την τελική έκθεση λοιπόν παρά στην ενδιάμεση έκθεση. Λοιπόν, το ε, ιστορικό Πώς ήρθε στην ενίσα αυτή η μελέτη, δηλαδή τον Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορίας, ε, που προήρθε και από τον Οργανισμό για την Άμυνα. Η ΕΝΙΣΑ ανέλαβε να επεξεργαστεί τις μελέτες αυτές. Έχουμε μία σύμβαση δηλαδή η οποία άρχισε να τρέχει πέρσι τον Οκτώβριο και εργαζόμεθα δηλαδή επί 6-7 μήνες στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα ήταν η μη ποσοτική προσέγγιση, δηλαδή χρησιμοποιήσαμε βιβλιογραφικά δεδομένα, ήταν τις διάφορες πολιτικές, ε, τα στοιχεία οικοδόμησης ικανοτήτων, τα προγράμματα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια η κοινή πολιτική ασφάλειας άμυνας. Μετά διατυπώσαμε ερωτηματολόγια, συντάξαμε ερωτηματολόγια που στείλαμε σε διαφόρους εμπειρογνώμονες ειδικού. Συμβουλευτήκαμε δηλαδή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για όλα αυτά τα στοιχεία και στο ΝΑΤΟ απευθυνθήκαμε, όπως είπε και η πρόεδρος πιο πριν, ε, επίσης κάναμε άλλες διαβουλεύσεις ε, εκτός ερωτηματολογίων με τους ειδικού. Αυτές είχαν τη μορφή συνεντεύξεων, είχαμε και επισκέψεις, πήγαμε στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, πήγαμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και άλλους ε, οργανισμούς και παράγοντες, έχω σχετική διαφάνεια και είχαμε και εσωτερικές συνεργασίες εντατικές. Η ομάδα που εκπροσωπούμε σήμερα αποτελείται από 6-7 ειδικού ε, στους κόλπους της Ενίσα που εργάστηκαν για τη μελέτη αυτή. Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες εκτός δηλαδή τον, του οργανισμού Ενίσα, όπως είπα πριν, κάναμε συζητήσεις με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Οργανισμό Άμυνας, συζητήσαμε και με τον ακαδημαϊκό χώρο, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από τη σχολή Λούι στην Ιταλία και ένα κέντρο έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συζητήσαμε πολύ και με συναδέλφους από τον ΝΑΤΟ, διάφορους τομείς, το κέντρο αριστείας που είναι στο Ταλίν, το CCDOE ε, τις επιχειρήσεις ε, συμμαχικής διοίκησης και την κεντρική διοίκηση του ΝΑΤΟ εδώ στις Βρυξέλλες. Και μιλήσαμε και με κάποιους ειδικού στον κυβερνοχώρο όπως το μέλλον στην Ελβετία. Τώρα, η θέση του προγράμματος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ε, Είμαστε στα τελικά στάδια, έχουμε ολοκληρώσει το 90% της μελέτης, αρχίσαμε τον Οκτώβριο, η τελική έκθεση θα υποβληθεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα και θα παρουσιαστεί στο Στρασβούργο, στην αρμόδια επιτροπή στις αρχές Απριλίου, στο Στρασβούργο αυτά. Μέχρι τώρα, τέλος Ιανουαρίου, όχι αρχές Ιανουαρίου δώσαμε την ενδιάμεση έκθεση, και η παρουσίαση της ενδιάμεσης έκθεσης γίνεται σήμερα. Επίσης έχουμε διατυπώσει και κάποιες ε, πολιτικές επιλογές που θα τις δείτε αργότερα, δηλαδή θα τις πούμε προς το τέλος της παρουσίασης αυτής και η τελική παρουσίαση θα γίνει στις 6 Απριλίου. Τώρα, το εύρος της μελέτης, αν δείτε αυτή την πυραμίδα από, πάν από κάτω προς τα πάνω, Έχουμε την θεκτικότητα των υποδομών, έχουμε τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και τέλος έχουμε πολύ συγκεκριμένα το πλαίσιο της ε, ΚΠΑ. Είδαμε την πυραμίδα για, με σκοπό να βελτιώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που καλύπτουν όλο το φάσμα, αρχίζοντας από τους κινδύνους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε όλους αυτούς τους τομείς. Η μελέτη, όπως ε, είπε η ΣΤΟΑ, καλύπτει τρεις θεματικούς τομείς, αρχίζοντας ε, από τα γενικά προς τα πιο ειδικά της ε, πολιτικής ασφάλειας άμυνας. Καταρχήν έχουμε τις πολιτικές προκλήσεις στον κυβερνοχώρο που εξετάσαμε τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη, το διεθνές επίπεδο, τις τεχνολογικές καινοτομίες, τις νέες τάσεις στην τεχνολογία που επηρεάζουν τον κυβερνοχώρο και ειδικότερα την ε, πολιτική ασφάλειας άμυνας. Είδαμε και τις συνεργασίες στα διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο ένωσης αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ο δεύτερος θεματικός τομέας καλύπτει την δημιουργία ικανοτήτων ε, για την ασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο γενικότερα. Είδαμε την κατάσταση των πραγμάτων σήμερα, τις διάφορες στρατηγικές, εθνικές και ενωσιακές στρατηγικές στον κυβερνοχώρο για την ασφάλεια. Ε, είδαμε δηλαδή τις ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που αποδίδονται και το ρόλο του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το ζήτημα της δημιουργίας ικανοτήτων. Ο τρίτος θεματικός, θεματικός τομέας είναι πιο στοχευμένος στην άμυνα στον κυβερνοχώρο και την ΚΑΠΑΑ. είδαμε το τοπίο απειλών σε σχέση με τις αποστολές ε, ε, σε αυτό το τομέα, ολοκλήρωση της άμυνας στον κυβερνοχώρο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τέλος τη συνεργασία Ένωσης ΜΑΤΟ. Πολιτικές επιλογές είδαμε έξι διαφορετικές κατηγορίες, ειδικότερα την ε, αντοχή, ισχύ στον κυβερνό πολιτική άμυνας, ε, ικανότητες στο, ε, πολιτικής ασφάλεια άμυνας, βιομηχανία, τεχνολογία και διεθνής πολιτική στον κυβερνόχώρο. χώρο. Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μας που ήταν μια γενική εισαγωγή στη μελέτη, το εύρος της, το ιστορικό της και τον τρόπο προσέγγισης από την πλευρά μας και τώρα ο Γιώργος Αντιχρίστος, ο συνάδελφός μου, θα μιλήσει περιεχόμενο για το περιεχόμενο και τα απορίσματα της μελέτης αυτής. Ευχαριστώ Παναγιώτη. Στα περίπου επόμενα 25 λεπτά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γενική εικόνα των πορισμάτων μας και να παρουσιάσω την αναλυτική μας δουλειά. Θα ξεκινήσαμε προσπαθώντας να χαρτογραφήσουμε τους στόχους που καθορίστηκαν από εκείνο που ανάθεσε το έργο και να καθορίσουμε το πλαίσιο. Έτσι ξεκινήσαμε και είδαμε ότι ο πρώτος και ο δεύτερος στόχος που μας ανετέθη είχε στόχο το πολιτικό και επίπεδο και ποια ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στατική προσέγγιση. Μετά εντοχή των υποδομών, θέλαμε να δούμε βασικά τι γίνεται στα κατώτερα στρώματα της δομής, της ΚΑΠΑΠΑ, τακτικό και τεχνικό επίπεδο. Και έχουμε τον ενδιάμεσο, τον επιχειρησιακό τομέα, την επιχειρησιακή στιβάδα, ε, που θεωρήσαμε ότι και εκεί θα έπρεπε να εστιαστούμε. Διότι θεωρούμε ότι η επιχειρησιακή αυτή πτυχή είναι πολύ σημαντική για την κυβερνοασφάλεια των αποστολών μας. Πώς συνεχίσαμε. Ξεκινήσαμε τους τρεις θεματικούς τομείς που περιέγραψε ο Παναγιώτης, προκλήσεις, δημιουργία ικανοτήτων και η πολιτική άμυνας και η κυβερνοασφάλεια και προσπαθήσαμε από εκεί να διατυπώσουμε ένα χάρτη προς την δημιουργία ικανοτήτων για την πολιτική μας. Και αυτός ο οδικός χάρτης καλύπτει και τα τρία στρώματα τα διοικητικά. Πολιτικά, στρατηγικά, επιχειρησιακά, τακτικά, τεχνικά επίπεδα. Ε, ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουμε ήταν μέσω μοντέλων. Θέλαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε κάποια μοντέλα που αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα για τη δημιουργία ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο και για τον έλεγχο προόδου και την οριμότητα των σχεδίων στο συγκεκριμένο μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Παγκόσμιο Κέντρο Κυβερνοασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί καθορίζεται η δημιουργία ικανοτήτων σε πέντε διαστάσεις που βλέπετε στη διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα, πολιτική κυβερνοασφαλείας και στρατηγικές. Δεύτερο, ενοτροπία, κουλτούρα και κοινωνία στον τομέα. Εκπαίδευση, κατάτηση και δεξιότητες, νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και μετά πρότυπα, οργάνωση και τεχνολογία. Όλη η δουλειά που κάναμε λοιπόν εστιάστηκε και βασίστηκε επί των πέντε διαστάσεων και προσπαθούμε στις προτάσεις μας να λάβουμε υπόψη αυτές τις πέντε διαστάσεις. Σε όλη μας τη δουλειά να το λάβουμε υπόψη και στα πορίσματα. Πάμε στο πρώτο τμήμα της μελέτης. Εντοπίσαμε εκεί τα βασικά προβλήματα για την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Εντοπίσαμε οκτώ προκλήσεις πολιτικής που θεωρούμε τις σημαντικότερες. Θα ξεκινήσω με το πρώτο στοιχείο ισορροπία μεταξύ των εξουσιών που υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ευθύνε. Αυτό που φεύγει και πέρα από το συγκεκριμένο τομέα τη ΚΑΠΑΠΑ είναι πιο ευρύ και σχετίζεται με το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κυριάρχων ε, κρατών και κάθε κράτο έχει προτεραιότητε πολιτικέ, στρατηγικέ για την κυβερνοασφάλεια. Απ' την άλλη βέβαια χρειάζεται και οργανωμένη προσέγγιση ειδικά από ΑΑ για την προστασία των υποδομών και των ανθρώπων που εκτελούν αποστολές εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το δεύτερο πρόβλημα είναι ο περίπλοκος, ε, το περίπλοκο σύνολο εντολών εντός των θεσμικών οργάνωσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διάφοροι θεσμοί που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια, διάφορες οργανώσεις, διάφορες υπηρεσίες και ούτω Άρα υπάρχει ανάγκη συνεκτικής προσεγγίσεως. Αυτό ήδη έχει δηλωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι χρειάζεται μια ε, συντονισμένη προσέγγιση για την κυβερνοασφάλεια στον τομέα που συζητούμε. Τρίτο πρόβλημα, η χρήση του κυβερνοχώρου στο, ε, στον πόλεμο και αν το διεθνές δίκαιο ε, εφαρμόζεται σε ένοπλες σειράξεις. Αυτό συζητείται ακόμα. Όσον αφορά το δυτικό ημισφαίριο υπάρχει συνένεση θα λέγα όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα του διεθνούς δικαίου στον κυβερνοχώρο, αλλά βέβαια χρειάζεται περισσότερη δουλειά να καθορίσουμε τις λεπτομέρειες και να ερμηνεύσουμε σωστά τα πάντα. Ε, αποκλίνουν οι απόψεις σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ δυτικού και ανατολικού ημισφαιρίου, όπως τα γνωρίζετε, η Κίνα και η Ρωσία έχουν διαφορετική άποψη από αυτού. Θεωρούν ότι ο κυβερνοχώρος ίσως να πετύχει ξεχωριστό νομικό πλαίσιο. Άρα εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δοθέτως, ο κυβερνοχώρος δεν έχει σύνορα. Το επόμενο πρόβλημα, πρόκληση. Οι ταχείες εξελίξεις όσον αφορά τις υβριδικές τεχνολογίες. Όλοι ακούμε για το διαδίκτυο των πραγμάτων, αλλά βλέπουμε και την χρήση υβριδικών τεχνολογιών στον πόλεμο. Άρα είναι σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Πώς θα ρυθμιστεί αυτή η όλη εξέλιξη και κυρίως στα πλαίσια που συζητάμε. Μετά, ταξονομία στον κυβερνοχώρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς, έχουμε διαφορετικούς ορισμούς όσον αφορά την ορολογία του κυβερνοχώρου. Νέες λέξεις αναδύονται καθημερινά όπως υβριδικός πόλεμος του κυβερνοχώρο, αντοχή του κυβερνοχώρου, ε, πρέπει να έχουμε συμφωνή γνώμη όσον αφορά την ορολογία του κυβερνοχώρου. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και να βασίσουμε τις προσπάθειές μας. Επόμενο πρόβλημα, αριθμός και επικοινομορφία των διαφόρων φορέων του κυβερνοχώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Όπως προανέφερα, κάθε χώρα έχει δική της άποψη για την κυβερνοασφάλεια. Άρα, Διαφορετικοί φορείς εμπλέκονται. Υπουργείο Δικαιοσύνη, Υπουργείο Άμυνα, Υπουργείο Εσωτερικών, δημόσιοι, ιδιωτικοί φορεί κέντρα αριστείας. Και πάνω από όλα αυτά έχουμε και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με την κυβέρνηση ασφάλεια. Η εναρμόνιση όλων των φορέων που συνεργάζονται κοινό όραμα είναι αρκετά δύσκολο. Επόμενο πρόβλημα. Η αλληλεπικάλυψη και πολιτικού τομέα. Οι απειλέ του κυβερνοχώρου στοχεύουν και τους δύο τομείς, στατιωτικό και πολιτικό. Άρα γίνονται πολλές προσπάθειες να υπάρξει καλύτερη άμυνα στον κυβερνοχώρο. Λόγω ελλείψεως συντονισμού και επικοινωνίας, πολύ συχνά βλέπουμε επικαλύψεις προσπαθειών και ίσως πατάλοι πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά για τη βελτίωση την γενικότερη τη ασφαλεία του κυβερνοχώρου. Μετά τέλο, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και να αναπτύξουμε πολιτική. Μιλάμε για απειλέ του κυβερνοχώρου την τελευταία δεκαετία λίγο πολύ και σε αυτή την περίοδο έπρεπε να καταλάβουμε τι είναι η απειλή, να δημιουργήσουμε οργανισμού και να συλλέξουμε στοιχεία, να μα βοηθήσουν τα στοιχεία αυτά, ούτω ώστε να αναπτύξουμε πολιτικέ και να τι προωθήσουμε. Δεν υπάρχει χρόνο να τα κάνουμε όλα αυτά. Και πέραν αυτού υπάρχει εγγενής δυσκολία ε, εντοπισμού των απειλών που είναι κάτι που δυσχεραίνει τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων. Προχωράμε τώρα. Από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για τη διαμόρφωση της σωστής πολιτικής και πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η καινοτομία στην τεχνολογία, η εξέλιξη στην τεχνολογία και πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε όλη αυτή την καινοτομία. Τα τελευταία χρόνια τι βλέπουμε. Ταχεία εξέλιξη σε δύο τομείς, σε δύο κατηγορίες θα έλεγα, στο διαδίκτυο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Είναι δύο τομείς που εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Απ' την άλλη βλέπουμε έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και προδιαγραφών του κυβερνοχώρου που θα βοηθούσαν να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνη για τη χρήση των ε, μέσων. Εκεί εστιαστήκαμε και σε αυτό να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτύξουμε προδιαγραφές και να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες βέβαια αφήνουν και ίχνος όσον αφορά ε, Τι αποστολές του πολιτικού και του τομέα στην ΚΕΠΑ. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης. Πάμε τώρα στην κατάσταση την παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άμυνα στον κυβερνοχώρο και το σχετικό πλαίσιο υφίστανται. Ε, εμπεριέχει ε, πέντε προτεραιότητες και 44 σημεία για να προωθηθούν για να αυξηθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, ερώτηση. Χρειαζόμαστε περισσότερα, αρκούν αυτά. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε σαν πρώτο βήμα να δούμε πού υπάρχουν κενά όσον αφορά το πλαίσιο. Επίσης να δώσουμε κάποιες απόψεις για επιχειρησιακό, τα διάφορα επίπεδα της ΚΕΠΑ. Επιχειρησιακό, τακτικό, τεχνικό, πολιτικό, στατικικό. Και πρέπει να παρακολουθούμε όλα αυτά τα, τις εξελίξεις, αυτά τα επίπεδα που προανέφερα. Τι κάναμε λοιπόν. Θέλαμε λοιπόν να αναλύσουμε και να χαρτογραφήσουμε στις πέντε διαστάσεις το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, του μοντέλου μας. Να εντοπίσουμε κενά, και να προτείνουμε συμπληρωματικά μέτρα για την ε, κυβερνοασφάλεια. Στα τρία επίπεδα της δίκησης της ΚΕΠΑ. Πάμε λοιπόν στην ΚΕΠΑ προσπαθώντας να δούμε ποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην ΚΕΠΑ. Πρώτα απ' όλα, τι βλέπουμε. Νέος τομέας συμπεριλαμβάνεται, ο κυβερνοχώρος. Γίνεται τομέας επιχειρήσεων. Έχει εντοπιστεί πολλά κράτη-μέλη στις εθνικές στρατηγικές του κυβέρνου χώρου και από άλλους διεθνείς φορείς, όπως το ΝΑΤΟ έχει εντοπιστεί. Άρα, έχουμε άλλο ένα τομέα επιχειρησιακό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό αποστολών και ΠΑΑ. Οι απειλές του κυβερνοχώρου μπορούν να παραχθούν σε αυτόν τον τομέα και να έχουν στόχο τον ίδιο τομέα, να έχουν στόχο άλλους επιχειρησιακούς τομείς ή ταυτόχρονα άλλοι τομείς μπορεί να αποτελούν απειλή για τον κυβερνοχώρο στην ΚΕΠΑ. Πάμε τώρα σε διοικητή επιχειρήσεων, σε μια αποστολή. Να μπούμε στο μυαλό του. Τι προσπαθεί να κάνει όταν εκτελεί την αποστολή του. Πρώτα απ' όλα θέλει να εντοπίσει το τοπίο των απειλών. Δηλαδή, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι κακοί. Και ποιοι δεν είμαστε σίγουροι αν είναι καλοί ή κακοί. Και βάσει αυτό αυτών, οι ηγέτες αυτοί, οι διοικητές, οι επιχειρησιακοί, έχουν χάρτες ανατομέα για να εντοπίσουν την απειλή για κάθε τομέα. Τι θέλουμε να κάνουμε. Να εισάγουμε τον τομέα τον καινούριο, τον κυβερνοχώρο και να εντοπίσουμε απειλές στον κυβερνοχώρο που θα μπορούσαν να βλάψουν τις αποστολές. Για να χειροτερέψει η κατάσταση, οι δεν είναι μόνο στο θέατρο των επιχειρήσεων που εμφανίζονται αλλά σε όλο τον κόσμο. Άρα αυτό για το διοικητή επιχειρήσεων είναι πολύ δύσκολο για να έχει μια σαφή εικόνα ποιο αποτελεί απειλή, από πού προέρχεται η απειλή ε, που στρέφεται κατά της ε, αποστολής του. Βλέποντας λοιπόν την εικόνα των αποστολών και πά, τώρα που μιλάμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε πολλές αποστολές οι οποίες είναι και αισθητικές και πολιτικές ή κοινέ αποστολές πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσης, οποιες ειναι και θετικέ και πολιτικες η κοινε αποστολες περα απο τα συνορα της ευρωπαικης πανω απο 5.000 άτομα α, ε, κινούνται εκεί και αυτοί οι άνθρωποι είτε είναι στρατιώτες είτε πολίτες χρειάζεται να έχουν ένα πλαίσιο κυβερνοασφάλειας, να τις προστατεύσουμε στον κυβερνοχώρο. Για αυτό το σκοπό έχουμε δύο παράλληλες δομές στην ΚΕΠΑ. Η μία για το στρατιωτικό τομέα, στρατιωτικές αποστολές και η άλλη για τις πολιτικές ε, αποστολές. Οι δύο δομές, οι διοικητικές δομές έχουν κοινό πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο Παρ' όλα αυτά έχουμε διαφορετικό διαφορετικές δομές σε επιχειρησιακό, τακτικό και τεχνικό επίπεδο, διαφορετικά αρχηγεία, κάποια αρχηγεία είναι ad hoc, έχουμε διαφορετικά αρχηγεία αποστολών. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και οι δύο δομές βρίσκονται στον ίδιο κυβερνοχώρο. Άρα η κυβερνοαπειλή μπορεί να επιτεθεί κατά της μίας ή της άλλης δομής ή κατά των δύο. Και επειδή η άμυνα στον κυβερνοχώρο είναι συλλογική προσπάθεια, άρα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο δομών, ούτω ώστε να έχουμε επαρκή, επαρκές επίπεδο άμυνας. Τώρα τι προτείνουμε εμείς. Προτείνουμε να υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την αξινόμηση των απειλών για το στρατιωτικό και τον πολιτικό τομέα και τι σχετικές αποστολέ στον κυβερνοχώρο, ε, έχουμε προτείνει λοιπόν αυτό εδώ, αυτή τη δομή που εδράζεται επί δύο πυλώνων. Ο πρώτος πυλώνας αφορά πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο και το επιχειρησιακό επίπεδο και δεύτερος πυλώνας επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση κατηγοριοποιούμε τις απειλές του κυβερνοχώρου για την ΚΕΠΑ σε τρία επίπεδα απειλής και έξι στιβάδες από τους ε, ερασιτέχνες hackers που το κάνει για διασκέδαση και πάμε μετά σε ομάδες που χρηματοδοτούνται από το κράτος και έχουν πολύ περισσότερες ικανότητες και δυνατότητες να προξενήσουν κάποιες ε, βλάβες. Και πέρα από αυτό προσπαθούμε να καθορίσουμε ένα εργαλείο που θεωρούμε ότι είναι χρησιμότατο για επιχειρησιακούς διοικητές, επιχειρησιακή χώρη αποκαλείται το εργαλείο, που είναι η απόσταση από τον επιχειρησιακό διοικητή μέχρι ε, το, κυβερνη, το πλήγμα στον κυβερνοχώρο. Έχουμε τρεις ορισμούς. Ε, εγγύς, μέσο, μέσης αποστάσεως, μακράς αποστάσεως. Στο κοντινό επίπεδο μπορεί να κινηθεί άμεσα ο διοικητής για να μυθεί. Μετά μέσο επίπεδο όπου η κυβερνοεπίθεση γίνεται στα δίκτυα και συστήματα που ελέγχονται και προστατεύονται από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μακρινές απειλές όπου Χρησιμοποιείται τα δίκτυα για αποστολέ ΚΠΑ και τα διαχειρίζονται ε, φορεί που δεν ανήκουν στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ανήκουν σε άλλε χώρε. Λοιπόν, τακτικό, ε, τεχνικό, επιχειρησιακό επίπεδο, σε αυτά τα επίπεδα, ε, έχει γίνει δουλειά από την ΕΝΗΣΑ όσον αφορά τον κυβερνοχώρο και την ταξινομία του κυβερνοχώρου. Και αυτή η δουλειά που έγινε εντοπίζει κυβερνοαπειλέ σε οκτώ κατηγορίε ταξινομή του κινδύνου. Οι δύο από τι κατηγορίε είναι αποκλειστικά του χώρου, του κυβερνοχώρου, Τι κατηγορίες είναι στο γενικότερο τομέα των πληροφοριών τη πληροφορική. οι άλλες απειλέ σχετίζονται με άλλους χώρου. Και αυτό είναι χρήσιμο για την ταξινόμηση και αξιολόγηση των απειλών του κυβερνοχώρου για την τεχνική στιβάδα και μετά αυτή η αξιολόγηση να προωθηθεί στο στην επιχειρησιακή στιβάδα, ώστε όλες οι πληροφορίες να συγχωνευτούν ούτω ώστε τελικά να διαμορφωθεί μια άποψη και μια αξιολόγηση σε επιχειρησιακό επίπεδο. Λοιπόν, τώρα για να επιλέξουμε πολιτικές, όπως προανέφερα, πρέπει να βάση το πλαίσιο πολιτικής για την κυβερνοάμυνα, να χατογραφήσουμε βάσει των πέντε ε, διαστάσεων του ε, μοντέλου που έχουμε για τη δημιουργία ικανοτήτων, εντοπίσουμε κενά και μετά να κινηθούμε με συμπροματικά μέτρα που προτείνουμε ότι πρέπει να ληφθούν ξεκινώντας από την πρώτη διάσταση. Θέλουμε να δούμε ποιε είναι οι επιλογέ πολιτικέ. Έχουμε τέσσερι κατηγορίε τη πολιτικέ. Ανταπόκριση στο επεισόδιο, προστασία κριτικών υποδομών, άμυνα του κυβερνοχώρου, αντοχή του κυβερνοχώρου. Για την όλη νοοτροπία και την κουλτούρα του κυβερνοχώρου θα πρέπει να διευρυνθεί η νοοτροπία στον αφορά να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, προστασία ταυτότητα, ε, κυβερνοέγκλημα, κοινωνικά μέσα, μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, πάνω από 55% των κυβερνοεπιθέσεων οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα, είναι η πλειοψηφία ανθρώπινο παράγοντα. Η τρίτη διάσταση εμπεριέχει δεξιότητες του κυβερνοχώρου και πώς εντάσσονται στις ε, ασκήσεις και επιχειρήσεις και πά, ε, νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια που αφορούν νομοθεσία, επιβολή του νόμου, προδιαγραφές, μέτρα και οδόμηση εμπιστοσύνης, διεθνή συνεργασία, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Μετά, τελευταία κατηγορία η αφορά την υιοθέτηση κοινών προδιαγραφών, ορολογίας, ε, ταξινόμησης των διαφόρων κινδύνων κλπ. Σημαντικό χρειάζεται να υπάρχει μια δομή μόνιμη άμυνας και πά εναντί των απειλών του και μετά θα πρέπει να υπάρξει αύξηση ικανοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών μελών. Τώρα συνοψίζοντας και ελπίζω να μην σας κούρασα υπερβολικά. Λοιπόν, πρώτο πόρισμα. Ο χώρος του κυβερνοχώρου δεν περιορίζεται στις ΚΕΠΑ. Ε, υπάρχουν επιτυχές και πολιτικές πέρα τη ΚΕΠΑ που πρέπει να εξεταστούν. Χρειάζεται συνοχή και οριμότητα που διαμορφώνεται μέσω σχηματισμού μοντέλων, όχι μόνο να καλύψουμε τα κενά, ώστε να παρακολουθούμε την οριμότητα και να δώσουμε τους κατάλληλους πόρους εκεί που χρειάζονται, να δημιουργηθεί ε, εμπιστοσύνη, αυτός είναι ο ανθρώπινος παράγων, ε, οργανωτικές αδυναμίες στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και τέλος κάτι εξίσου σημαντικό, η ένταξη ε, του κυβερνοχώρου στις επιχειρήσεις ΚΕΠΑ και στον πολιτικό και σε τομέα και εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και αν έχετε τυχόν ερωτήσεις με τα χαράς να απαντήσω. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για αυτήν την ε, πληρέστατη παρουσίαση της μελέτης. Ο κύριος Γκάλερ καταρχάς έχει το λόγο. Θα, ζητήσω, θα μιλήσω γερμανικά, λέει ο μιλητής. Καταρχήν, συγγνώμη, ε, έπρεπε να πάω παράλληλα και να μιλήσω και σε άλλη συνεδρίαση και δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Αλλά το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης το παρακολούθησα και νομίζω ότι εκεί είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε. Ε, τώρα, το, στον κυβερνοχώρο ε, έγινε αναφορά στο δίκαιο ένοπλων ε, συγκρούσεων. Εδώ πρέπει να πάρουμε σαφή θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γιατί αυτό πρέπει να εφαρμοστεί αν ας πούμε ε, κλείσω την παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος σε μια χώρα δεν είναι σαν δήλωση πολέμου, δεν είναι σαν να ρίξω βόμβα ε, ή αν όπως αν βομβαρδίσω το, τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, αν θέλω δηλαδή να παραλύσει ο αντίπαλος, μπορεί να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να την δούμε και σε νομικό επίπεδο ε, και να δούμε το δίκαιο του πολέμου σε αυτά τα πλαίσια. Υπάρχει βέβαια και ένα δίλημα έχω, γενικά στη συνεργασία στον κυβερνοχώρο, ότι δηλαδή αν θέλαμε να γενικά να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, τότε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποκαλύψει τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του. Αυτό μπορεί να μην γίνεται ούτε στους κόλπους μιας χώρας, πόσο μάλλον απέναντι σε ένα άλλο κράτος μέλος. Η στάση αυτών των αρχών είναι κάπως, δηλαδή μπορεί να ε, αντιμετωπίζουν εχθρικά και τον υποτιθέμενο φίλο, καμιά φορά περισσότερο και από τον αντικειμενικό εχθρό. Ίσως λοιπόν ε, να πρέπει να, το, να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα, ότι δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει ε, άνοιγμα. Για τις προκλήσεις της ΚΕΠΑ, εδώ εστιάζουμε περισσότερο στις αποστολές, και θα ήθελα να ρωτήσω αν όντως ε, κάποιος που συμμετέχει σε μια αποστολή της ΚΕΠΑΑ φέρει τα, το δικό του συναφές υλικό, ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι ήδη μολυσμένο με ιούς. Εμείς ε, στα πλαίσια των αποστολών μας, στις επικοινωνίες, σε τομέα δηλαδή σχετικό με τον κυβερνοχώρο, θέλουμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Πώς θα το αποφύγουμε. Μήπως ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ε, φτιάχνουμε από κοινού υλικό αυτό και να το διαφυλάσσουμε ε, για τις αποστολές αν γίνουν. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα έχει διασφαλιστεί η καλή του κατάσταση, θα προστατεύεται και έτσι θα έχουμε κάποιες εγγυήσει ότι δεν θα υπάρξει εξωτερική μόλυνση κατά τη διάρκεια της αποστολής. Συμβαίνει αυτό ή υπάρχει κάποια αξιόπιστη προοπτική να καταλήξουμε εκεί ούτως ώστε οι αποστολές μας να έχουν προφυλαγμένο και προστατευμένο άρα και απρόσβλητο υλικό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σαφχάουζερα. Ναι, Πρόεδρε, δεν θα με ακρηγορήσω. Η εμπειρία μου, γιατί έχω εργαστεί στο στρατιωτικό τομέα, είναι ότι αν δεν ελέγχουμε απολύτως τις διαδικασίες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ασφάλεια. Δηλαδή, από το λογισμικό, στο hardware, στο router, στα ηλεκτρονικά chip, στα συστήματα διαβίβασης, ξεκινώντας από το chip, αν δεν τα ελέγχουμε όλα αυτά δεν μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι. Ο κατασκευαστής του τσιπ δεν μπορεί να γνωρίζει απολύτως αν ένα συγκεκριμένο τσιπ μπορεί να προσβληθεί ή όχι. Και εδώ μιλάω για επικυριαρχία ή δυνατότητα αμήνης και ελέγχου επί του λογισμικού, γιατί το hardware στην ουσία υπάγεται στο λογισμικό υπό μία έννοια. Δηλαδή, ποιος μπορεί να προσβάλλει το Windows 10, το λειτουργικό σύστημα του Windows 10, χωρίς να σας ρωτήσει καν. Η μόνη εταιρεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που κατασκευάζει τσίπ ηλεκτρονικά σήμερα δεν ξέρει αν θα επιβιώσει. Χρειαζόμαστε 20 με 30 δισεκατομμύρια επενδύσεις για να είναι απλώς, για να παρακολουθεί απλώς τους υπόλοιπους παγκοσμίους ανταγωνιστές της που είναι πέντε. Αυτό είναι αφενός πολύ σημαντικό λοιπόν. Αφετέρου, όλες οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Προς το παρόν έχουμε δει ότι ήταν αναγκαστικά οι Ρώσοι που έκανα τις επιθέσεις ή κατασκοπία. Βέβαια, οι γερμανικές και γαλλικές ηγεσίε δεν μιλούν πλέον, πολιτικές ηγεσίε δεν μιλούν πλέον γι' αυτό. Αλλά έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα στο επίπεδο αυτό και επίσης καθότι εγώ συμμετείχα στις ερωτήσεις αυτές αυτό που θα μπορούσαμε να, που, να κάνουμε, όπως οι Αμερικανοί που έχουν ένα κέντρο, δεν θυμάμαι σε ποια πρεσβεία, πρόσφατα αποκαλύφθηκε, θα μπορούσε κανείς να κάνει μια επίθεση να φαίνεται ότι ε, προέρχεται από τους Ρώσους. Να την φτιάξει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι οι Ρώσοι την έκαναν. Όλα αυτά είναι αρκετά περίπλοκα λοιπόν. Επομένως, ο μόνος τρόπος να ελέγξουμε, να αμυνθούμε είναι να ελέγχουμε απολύτως και το λογισμικό και τον ε, εξοπλισμό, το hardware. Γιατί αν το υλικό που έχουμε ελέγχεται από άλλους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αμυνθούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ είχα μια σειρά από ερωτήσεις. Υποθέτω ότι θα έχετε κάνει μια ανάλυση επί τη βάση τη οποία κάνατε την έκθεση αυτή. επομένω, ποιοι είναι οι πιο, οι πιο τυπικές μορφές επιθέσεων κυβερνοχώρου αφενός, Ποιε είναι. Επίσης, σε τι επίπεδο γίνεται, σε υψηλό επίπεδο, σε χαμηλό. Εγνωρίζουμε ότι οι εθνικές στρατιωτικές ε, ε, δυνάμεις ε, επικεντρώνονται περισσότερο σε απειλές στρατιωτικού επίπεδου των πολεμικών επιχειρήσεων. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ενέχονται σε θέματα αμήνης κυβερνοχώρου. Αλλά ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει κρούσματα παρακολούθησης κατά και μελών του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ηγεσιών. Και μάλιστα ίσως και από εντός εγωγικών φίλους. Μάλιστα σε ευχαριστώ κύριο Μπούχνα μια σύντομη παρατήρηση. Ακούμε και το είδα ε, ε, ε, και εγώ αυτό και σας ρωτώ. Υπάρχει εντωμεταξύ Ευρωπαϊκό Κέντρο το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την αντικατασκοπία γιατί ακούσαμε περιστατικά, τα ανέφερε και ο κύριος Γκάλερ, συστηματικής διείσδυσης σε ορισμένα προγράμματα. Ε, για τη λήψη στοιχείων. Δηλαδή εδώ βρίσκεται σε αδυναμία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνει τίποτε. Δηλαδή ε, υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιος είναι. Σας, Σας ευχαριστώ. Έχω κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών. Επομένως, κύριοι, ο λόγος δικός σας. Μάλιστα, πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση. Την πρώτη παρατήρηση. Σχετικά με την ανάγκη εμπιστοσύνη. Συμφωνούμε ότι πράγματι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και μάλιστα το υπογραμμίζουμε στη μελέτη. Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης είναι μια διαδικασία συνεχιζόμενη. Προτείνουμε κάποια μέτρα λοιπόν ε, εντός της μελέτης που μπορούν να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη αλλά ξαναλέω είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίζεται δεν μπορεί να διακοπεί, δεν μπορούμε να το παγώσουμε σε μια χρονική στιγμή. Τώρα, για τον κοινό εξοπλισμό της αποστολές ΚΕΠΑ. Αυτό είναι κάτι που δεν υφίσταται. Πρόσφατα ήμασταν σε μια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης που έχει αρχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή αλλά δεν έχουμε ακόμη κάτι τέτοιο. Πράγματι το να έχει κανείς κοινά εργαλεία είναι πολύ σημαντικό αλλά θα μπορούσε να πει κανείς κάτι περισσότερο. Όχι μόνο κοινά εργαλεία, να έχει κοινή κεντρική διοίκηση ικανότητας που να μπορεί να υποστηρίζει τις πτυχές του κυβερνοχώρου της κάθε επιχείρησης ή αποστολής. Για, για τις κατασκευές των ηλεκτρονικών τσίπ ε, είναι κάτι, ένα πρόβλημα πάρα πολύ γνωστό. Η όλη, το όλο θέμα της υποδομής IT ε, δεν έχει επιληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, το πιο ισχυρό μας επιχείρημα εδώ, η θέση, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει, να υποστηρίξει οπωσδήποτε την Ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρον, ε, πληροφορίας ηλεκτρονικής, της ε, κοινωνίας της πληροφορίας, IT τέλο πάντων. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο στον κλάδο, στη βιομηχανία, για να ενδυναμωθεί συνολικά η βιομηχανία. Οι τεχνολογικές διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές και λέω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το ευρωπαϊκό κλάδο, αλλά θεωρούμε ότι τα προβλήματα κάθε αυτά δεν είναι τεχνολογικής φύσεως. Τα πιο δύσκολα είναι είτε οργανωτικής φύσεως είτε νομικής. Δηλαδή είναι και αυτές τις πτυχές που πρέπει να εξετάσει κανείς ως πτυχές που αφορούν άμεσα στην πολιτική. Για τις επιθέσεις ε, στον κυβερνοχώρο που μπορούν να προέρχονται και από συμμάχους. Εδώ τα σημαντικά σημεία είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο συνάδελφος ίσως να πει περισσότερα, για τις δε πιο κοινέ, πιο συνήθεις επιθέσεις, είχαμε κάνει μια χαρτογράφηση των απειλών, βλέπετε αυτόν τον πίνακα, που είναι στο πλάι. Είναι μια δουλειά που κάνουμε κάθε χρόνο και ως ανεξάρτητος οργανισμός είμαστε αντικειμενικοί στα όσα τοποθετούμε στον πίνακα αυτό. Έχουμε τις δύο στήλες με τις ε, ισχύουσες απειλές για το 2015 και για το 2016. και με την τάση Προ τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την σημασία, τη σοβαρότητα τη απειλή. Μιλάμε για malware, ε, επιθέσεις ε, άρνησης ε, παροχής υπηρεσίας, μπλοκαρίσματος της ροής των πληροφοριών και διάφορες άλλες. τα δημοσιεύουμε αυτά κάθε χρόνο και ονομάζονται οι εκθέσεις αυτές ENISA Threat Landscape, δηλαδή η χαρτογράφηση της απειλής περίπου, και για την ύπαρξη ενός κέντρου που θα μπορούσε να χειρίζεται θέματα κατασκοπίας ή παρακολουθήσεων, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, εξ όσων εγώ γνωρίζω. Και να προσθέσει ο Γιώργος κάποια πράγματα, ευχαριστώ. Κάποια ακόμα σχόλια για τα διάφορα πολύ ενδιαφέροντα που αναφέρατε. Για το διεθνές δίκαιο είναι μεγάλο θέμα αυτό. Καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουμε. Μία προσέγγιση θα ήταν να έχουμε πιο συνεπείς στρατηγικές ε, για τον κυβερνοχώρο μεταξύ των κρατών μελών και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεισφέρουμε συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ε, υιοθέτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνη, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό που είναι όμως καθόλου εύκολο. Υπάρχει τεράστια διχογνωμία όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά συνολικά θα έλεγα στο δυτικό ημισφαίριο. Για το δυναμικό για την ε, ευρωπαϊκή ικανότητα ε, πρέπει πράγματι να έχουμε εχέγγυα για το τι είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσει κανείς. Για τα είδη των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ο Παναγιώτης σας μίλησε για την, ε, τις χαρτογραφίες της αιτήσεις της ΕΝΗΣΑ, αλλά μπορώ να σας πω επίσης ότι στη μελέτη έχουμε τρεις μελέτες τύπου περίπτωσης με σενάρια και τι θα συνέβαινε, ποιο θα ήταν ο αντίκτυπος υπό το κάθε σενάριο. Θα μπορούσαμε να έχουμε επιθέσεις κυβερνοχώρου και στα τρία επίπεδα διακυβέρνηση που παρουσιάσαμε. Όπως λέμε, στη μελέτη, είμαι βέβαιος ότι θα έχετε ακούσει για τις πρόσφατες ε, επιθέσεις ε, στην Ουκρανία, η επιθέσεις κυβερνοχώρου. Είναι ένα κομμάτι της ψυχολογικής προσπάθειας επίθεσης και στοχοθετεί τις υποδομές κρίσιμης σημασίας. Μπορεί να γίνει λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Θα μπορούσε να γίνει αυτό κατά μόνο στρατιωτικών ή αμυντικών συστημάτων. Και παρουσιάζουμε και μία περίπτωση πριν από 10 χρόνια όπου μία χώρα χρησιμοποίησε συστήματα κυβερνοχώρου για να μπλοκάρει ραντάρ. Και να επιχειρήσει λοιπόν αεροπορικές επιθέσεις χωρίς να έχει ανεχρευτεί. Επομένως, εδώ μιλούμε για στοχοθέτηση στρατιωτικών υποδομών. Άλλες επιθέσεις θα μπορούσαν να στοχοθετούν την ίδια την αποστολή ΚΕΠΑ. Είχαμε στην Λατινική Αμερική επίθεση επί 10 χρόνια μέρος ε, οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητα. που σχετιζόταν και με το πολιτικό επίπεδο ή μάλλον έπληκε το πολιτικό ε, επίπεδο, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει και την αξιοπιστία της αποστολής ή και της χώρας που την φιλοξενεί. Πρέπει λοιπόν να δει κανείς τις επιθέσεις αυτές του κυβερνοχώρου σε κάθε επίπεδο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό μόνο σε ένα επίπεδο ή θα μπορούσε να συντονίζεται σε διάφορα επίπεδα. Για την τελευταία ερώτηση που κάνατε για την ανάπτυξη του δυναμικού έχουμε το, το κέντρο πληροφοριών ε, ε της ΙΕΔ αλλά συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι δεν έχουμε κάποιο αφιερωμένο κέντρο που θα το με παρακολουθήσεις ή θέματα ε, προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν ζητεί άλλο τον λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δύο κυρίους για την ε, ε, πλήρη αυτή ενημέρωση, για τη μελέτη ενίσα ε, βεβαίως θα μείνουμε σε επαφή αφού η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα θέμα που θα το αξιολογήσουμε και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και από κοινού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτό το διήμερο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ενδελεχείς ε, διαβουλεύσεις. Ελπίζω ότι η μερίσια διάταξη είχε ενδιαφέρον για όλους σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους διερμηνείς για τη σκληρή δουλειά, τη γραμματεία επίσης. Στα διάφορα δεν έχουμε τίποτε, γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Η προσεχή συνεδρίαση είναι στις 11 Απριλίου και 12 Απριλίου. Ε, ελπίζω να σας καλωσορίσω εκεί. Ευχαριστώ.